Man sollte normalerweise, liebe Kolleginnen Kollegen, nicht die bestrafen, die Δεν θα περιμένουμε παραπάνω. Όποιο δεν είναι στην ώρα του, νομίζω ότι δεν μπορούμε να τον περιμένουμε παραπάνω. Θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω την ομάδα που εργάζεται για την ε, κυβέρνηση της Ταϊβάν. Είναι εδώ μαζί μας και θα παρακολουθήσουν την σημερινή μας ε, συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και ελπίζω να περάσετε μια ευχάριστη συνεδρίαση εδώ μαζί μας και να μάθετε κάποια πράγματα. Πριν συνεχίσουμε με το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η παρουσίαση της ε, έκθεσης από την Rand Europe, της μελέτης μάλλον, για την εκπαίδευση και την νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικές προκλήσεις, ε, μελλοντικές προοπτικές για θέματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά θέματα, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, European Affairs και το PPMI. Θα ήθελα καταρχήν να ακούσουμε μία σύντομη παρουσίαση για το αρμόδιο τμήμα να μας ε, εξηγήσετε πώς ακριβώς στηρίζετε τις εργασίες από το Policy Department, τις εργασίες της σημερινής μας, αλλά και τις μελλοντικές μας εργασίες εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού. Κύριε Λίτσελμαν, θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Χαίρομαι που ήρθατε σήμερα εδώ και έχετε το λόγο για να μας κάνετε μια σύντομη παρατήρηση. Βεβαίως, οι ερωτήσεις μπορούν να γίνουν και κατευθείαν στον κύριο Λίτσελμαν, αλλά μην ξεχνάτε ότι σήμερα είμαστε εδώ κυρίως για να παρουσιάσουμε αυτήν την μελέτη που έκανε η Rand Europe. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ στις εργασίες, λέει ο κ. Λίτλμαν, του Policy Department Β. Αυτό δημιουργήθηκε το 2004 με σκοπό να στηρίξουμε τη γραμματιακή εργασία της Επιτροπής. Όλες οι επιτροπές, αν θέλετε, συνδέονται με ένα συγκεκριμένο τέτοιο τμήμα Policy Department. Είναι κάτι που, όπως βλέπετε, και στη διαφάνεια έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμάς, αρμοδιότητά μας είναι οι μεταφορές, η Ρέτζη, η ΠΕΣ και βεβαίως η Επιτροπή Πολιτισμού, η δική σας Επιτροπή. Υποστηρίζουμε με πραγματογνωμοσύνη όχι ε, ατομικά κάποια μέλη του Κοινοβουλίου ή κάποια μέλη των Επιτροπών, αλλά συνολικά ε, τις ε, Επιτροπές ε, και τα διάφορα θεσμικά όργανα. Βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει μετά από συγκεκριμένες αιτήσει των βουλευτών, των μελών της Επιτροπής με σκοπό να βοηθήσουμε την λήψη πολιτικών αποφάσεων. Παραδείγματο χάρη κάποια νομικά, τεχνικά ή οικονομικά θέματα μπορεί να διευκρινιστούν, να αποσαφινιστούν μετά από τις δικές μας μελέτες, θέματα που αφορούν επίσης την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, θέματα που αφορούν δημοσιονομική πολιτική, Έχουμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι καλύπτουν όλα τα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική. Υποβάλλουμε λοιπόν μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, οι οποίες ουσιαστικά χαρακτηρίζονται από την δράση που πρέπει να ακολουθήσει. Υποβάλλουμε συστάσεις, εναλλακτικά σενάρια, κάτι που θα μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη μας πάντα τις στρατηγικές προτεραιότητες όπως τις έχετε εσείς καθορίσει. Για επίσης κάποια θέματα που είναι πολύ πιο λεπτά μας αφορά δηλαδή η δική σας ε, θέση προτεραιοτήτων με σκοπό να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, να σας βοηθήσουμε να τηρήσετε τους κανόνες, παραδείγματος χάρη μιας υποβολής προτάσεων ενός διαγωνισμού. Έχουμε συγκεκριμένες διαδικασίες και βεβαίως ε, οι περισσότεροι που εργάζονται στο δικό μας ε, Policy Department είναι εμπειρογνώμονες, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και βεβαίως ερχόμαστε εδώ, σας παρουσιάζουμε τις εκθέσεις ε, και ανταλλάσσουμε απόψεις μαζί σας. Βλέπετε εδώ τις παρουσιάσεις που κάνουμε, μελέτες, εις βάθος μελέτες, αλλά και μικρές ενημερωτικές παρουσιάσεις. Οι μελέτες μας προετοιμάζονται και δημοσιεύονται στα αγγλικά. Έχουμε πολύ περιορισμένες δυνατότητες ε, μετάφρασης και βεβαίως δίνουμε προτεραιότητα όταν πρέπει να γίνει μετάφραση σε κάποια νομοθετικά κείμενα. Οι μελέτες μας πολλές φορές ε, μπορεί να μας ζητηθεί να μεταφραστούν, αλλά αυτό γίνεται σε μία ή δύο γλώσσες. Οργανώνουμε επίσης ε, εργαστήρια και κάνουμε και εξαιρετικές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρουσιάσεις εκτός των θεσμικών οργάνων. Αυτά όλα πρέπει να σας πω τα καλύπτουν οι συνάδελφοι. Έχουμε δύο συναδέλφους, τις κυρίες Ίσκα και Ήρια, οι οποίες αφιερώνουν το χρόνο τους ε, για την Επιτροπή Πολιτισμού, τη δική σας ε, ε, Επιτροπή. Οι διαδικασίες ε, δημόσιων συμβάσεων, όπως βλέπετε εδώ, η διαδικασία αυτή είναι θεσμοθετημένη. Το μειονέκτημα αυτών των διαδικασιών είναι ότι ξεκινάνε πάντα από μια συγκεκριμένη απόφαση της δικής σας Επιτροπής, παραδείγματος χάρη, για να αναλάβουμε μια αποστολή, μια μελέτη Ξεκινάμε με κάποιους μήνες στους οποίους τεκμηριώνουμε την έρευνά μας και ακολουθεί ο έλεγχος της ποιότητας και ενδεχομένως η μετάφραση. Και βλέπετε και το χρονοδιάγραμμα. 4 με 12 μήνες, 4,5 με 12 μήνες είναι ο μέσος όρος. Όλα αυτά τα κείμενα, όλες αυτές οι μελέτες ε, είναι δημόσιες στο ίντρανετ, αλλά και στο διαδίκτυο. Μπορούμε να παρέχουμε και περισσότερες πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα και βεβαίως υπάρχουν και σε έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη. Πολύ σύντομα θέλω να σας υπενθυμίσω τι κάναμε στην τελευταία θητεία, πώς συνεργαστήκαμε πάνω από 40 μελέτες, κινητικότητα των καλλιτεχνών, επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού, το Erasmus Plus και η ε, μελέτη μας για την ενιαία αγορά στον τομέα του πολιτισμού. Διοργανώσαμε επίσης πέντε εργαστήρια, εργαστήρια που αφορούν το ψηφιακό κόσμο, τις νέες τεχνολογίες, και αυτές τις μελέτες τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει και θα παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον. Επίσης, έχουμε και όλες τις μελάτες τις οποίες θα πρέπει να προετοιμάσουμε εν ώψη του 2020. Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό και έξυπνο τρόπο τα κονδύλια που διαθέτουμε, στηριζόμενοι πάντα και ακολουθώντας τις ε, προτεραιότητες που θέτουν οι επιτροπές για τις οποίες εργαζόμαστε. Περιμένουμε από εσά και από τις πολιτικές ομάδες συγκεκριμένη ενημέρωση, feedback, έτσι ώστε να μας κατευθύνετε προς τους τομείς αυτούς που θεωρείτε εσείς εξαιρετικά σημαντικούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λίτσαμαν, λέει η Πρόεδρος. Θεωρώ ότι η στήριξή σας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για μας, για την δουλειά μας και ελπίζω ότι αυτή η εξαιρετική συνεργασία, η στενή συνεργασία θα συνεχιστεί και στην επόμενη θητεία. Θέλει κάποιος πριν περάσουμε στη μελέτη, στις μελέτες, να πάρει το λόγο, να κάνει ερώτηση προς τον κύριο Λίτσελμαν. Όχι. Χαίρομαι πάντως γιατί είπατε είσαστε στη διάθεσή μας για περαιτέρω συνεργασία και μελέτες. Και θα περάσουμε τώρα στη μελέτη που ζητήσαμε στην προηγούμενη θητεία, στις δύο μελέτες. Σήμερα θα πρέπει να στοχεύσουμε τις δύο πολύ σημαντικές προτεραιότητες θα δώσω το λόγο στην Αξέλ Δελβό και την Φέι Ντάνκερλι από την RAND Europe. Το θέμα μας είναι η εκπαίδευση και οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα σενάρια που έχετε να μας παρουσιάσετε, οι επιπτώσεις τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε και να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ και τις δύο. Σας δίνω το λόγο. Ε, καλό θα ήταν να μην ξεπεράσετε τα 15 λεπτά. Έχετε το λόγο. Thank you. Good afternoon and thank you Γεια σας, ευχαριστώ που μας καλέσατε για να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης θα σας εξηγήσω ποια είναι η εργασία που κάνουμε, για ποιο λόγο κάνουμε αυτό που κάνουμε, με ποιο τρόπο και ποια είναι τα ευρήματα. Χρησιμοποίησαμε μία άδοξη προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική εκπαίδευση και νεολαία. Θα ακούσετε για να γίνεται λόγος για κάποια σενάρια για πρώτη φορά σήμερα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο και πώς χρησιμοποίησαμε αυτά τα σενάρια. Ξέρουμε ότι η εκπαίδευση και η πολιτική για την νεολαία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον. Οι διάφορες μελέτες μπορούν να μας βοηθήσουν για να δούμε περίπου πώς, με τι θα μοιάζει το μέλλον και ποιες είναι και εναλλακτικέ λύσει σε θέματα παιδεία. Ο στόχο λοιπόν αυτή τη μελέτη είναι να βοηθήσει εσά, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να καταλάβετε πώ ε, λαμβάνετε υπόψει για το μέλλον. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε διάφορες προσεγγίσεις, κάποια σενάριο για να μπορέσουμε να απεικονίσουμε πώς προβλέπετε ότι θα γίνουν και διάφορες αλλαγές στα 10-15 επόμενα χρόνια, όχι μόνο σε θέματα παιδείας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ε, τις τεχνολογικές εξελίξεις, κοινωνικο, κοινωνικο, οικονομικά κριτήρια και αν δούμε ποιος, είναι ο αντίκτυπος της διάφορες εναλλακτικές λύσεις, θα καταλάβετε τι κάνουμε. Πώς προχωρήσαμε. Πρώτα απ' όλα κάναμε αναθεώρηση των διαφόρων εγγράφων που διαθέτουμε για τις πολιτικές Ευρωπαϊκές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη διάφορους δείκτες το ΑΕΠ. Οι αλλαγές στο ΑΕΠ μπορούν να επηρεάσουν τα θέματα τα εκπαιδευτικά. Δεύτερον, ήρθαμε και σε επαφή με διάφορους εμπειρογνώμονες. Βασιστήκαμε σε διάφορες ε, προσεγγίσεις, κάναμε διάφορες προβολές. Πήραμε εδώ ως δείκτη της προβλέψεις Μπορεί το ΑΕΠ να μείνει στάσιμο, να αυξηθεί, να μεταβληθεί, πράγμα το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον. Αυτό είναι μια προβολή. Επίσης είδαμε σε ποιο μέτρο οι δύο αυτές προβολές είναι συνεχτικές μεταξύ τους. Αν επανέλθω στο πράγμα του ΑΕΠ, μπορείτε να φανταστείτε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει αύξηση ε, του ΑΕΠ, αλλά στασιμότητα στα θέματα Αυτά λοιπόν είναι κάποια δυνατά σενάρια για το μέλλον. Μετά είδαμε ποιες ήταν οι πολιτικές ενδεχομένως σε σχέση με κάποια σενάρια τα οποία δεν ήταν πραγματικά, κάποια ήταν ελευθερισμένα, κάποια οικονομικά. Για να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις πολιτικής. Πρώτα απ' όλα εντοπίσαμε πέντε ε, εναλλακτικές Εξετάσαμε πρώτα απ' όλα τις εναλλακτικές λύσεις στην πολιτική όποιο και να είναι το μέλλον, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Λάβαμε υπόψη διάφορα σενάρια κοινωνικο-οικονομικά, ε, λάβαμε υπόψη διάφορες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δεν είναι, ε, αποκλείουν μεν τις δε. Θα μπορούσαν λοιπόν και τα πέντε, η πέντε αυτές εναλλακτικές λύσεις να είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους και να εφαρμοστούν όλα. Η πρώτη είναι η μάθηση επικεντρωμένη στους φοιτητές με ευέλικτο τρόπο. Δεύτερη, συμπεριληπτική μάθηση της ψηφιοποίησης, δηλαδή όλοι συμπεριλαμβάνονται στη νέα εποχή της ε, ψηφιοποίησης. from education are further excluded. Τρίτη εναλλακτική λύση είναι να επενδύσουμε το συντομότερο δυνατό σε θέματα ε, εκπαίδευσης ώστε να μην διονυστούν κάποια ε, θέματα τα οποία θεωρούμε ότι έχουν αρνητικό χαρακτήρα. Και πέμπτον, θέλουμε όλοι αύριο οι πολίτες, όποιο και να είναι το μέλλον, να συμμετέχουν ισότιμα στις κοινωνίες τις οποίες ζουν. Επίσης, Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, στις αλλαγές, δεδομένου ότι είναι κλειδί για την εκπαίδευση των νέων. Τώρα επανερχόμαστε στα διάφορα σενάρια. Τα τέσσερα, τα οποία αναπτύξαμε. Έχουμε τέσσερα σενάρια εντελώς διαφορετικά σε σχέση με διάφορα τομείς κλειδιά που δεν είναι μόνο αυτό της εκπαίδευσης αλλά και σοσιοοικονομική. Και θα σας παρουσιάσουμε κάθε σενάριο χωριστά για να δούμε κατά πόσον συνάδουν με τις πολιτικές επιλογές και προσεγγίσεις που ε, θα ακολουθήσουμε. Το πρώτο λέγεται κατακαιρματισμένη Ευρώπη, ευθυγραμμισμένη Ευρώπη, η Ευρώπη με τα κρύα πόδια και η Ευρώπη στρουθοκάμιλος, που στρουθοκαμιλίζει. Ας δούμε το πρώτο σενάριο. Κατακαιρματισμένη Ευρώπη. Εδώ το σύστημα, τα εκπαιδευτικά δεν μπόρεσαν να ετοιμάσουν νέους ανθρώπους για να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας στη σημερινή ψηφιοποιημένη ε, εποχή μας. Κάποιοι μόνο είναι προετοιμασμένοι. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι τέτοιου είδους πολιτικές θα οδηγήσουν σε τέτοιο ε, αποτελέσματα. Δεύτερο σενάριο. Συγγραμμισμένη Ευρώπη. Πρώτη προτεραιότητα, η σωστή εκπαίδευση. Για όλους. Όλους όσους φύστανται την μαθησιακή διαδικασία. Και η πάρα πολύ καλός συνδυασμός μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και των αναγκών της αγοράς. Το τρίτο σενάριο. Κρυώνουν τα πόδια της Ευρώπης. Εδώ η ψηφιοποίηση έχει θετικό πρόσημο ε, στην οικονομία, αλλά υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και πολλούς νέους τους απασχολεί το μέλλον. Έχουμε το πρόβλημα μεταξύ των, ε, της Ευρώπης της παλιάς γενιάς και το πώς πρέπει να προετοιμάσουμε για την ψηφιοποιημένη και τη μοντέρνα και γεννή τους νέους. Εδώ λοιπόν όλοι επηρεάζονται από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, αλλά η, το, η αντίδραση, η ανταπόκριση στους καινούργιες τεχνολογίες και στην ψηφιοποίηση είναι πολύ αργότερη. Τέταρτο σενάριο. Η Ευρώπη στουρθοκαμιλίζει. Δηλαδή, οι πολιτικές της παιδείας ε, έχουν, ε, προχωρούν ως έχουν, δίδονται κονδύλια, αλλά είναι κάπως στεγανά η εκπαίδευση. Φαίνεται λοιπόν ότι μακροπρόθεσμα ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι το καλύτερο. Έχουμε λοιπόν μία πολύ περιορισμένη εμβέλεια εφαρμογή των σενάριων που παρουσιάσαμε. Βλέπετε λοιπόν πως κάθε εναλλακτική λύση θα μπορούσε να συνάδει με τέσσερα σενάρια προβλέψουμε, προβλέπουμε για την Ευρώπη για το μέλλον. Δεν λέει σε εσάς που είστε ε, ευρωβουλευτές τι πρέπει να κάνετε, αλλά θέλει να καταδείξει πώς με τις αποφάσεις μπορείτε να επηρεάσετε τα αυριανά σενάρια την Ευρώπη. Αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε με τις ε, πολιτικές εκπαίδευσης και όλες τις πολιτικές για τους νέους είναι να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχείς πολιτικές και βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται και από αυτά τα οποία θέλετε εσείς ως Επιτροπή να επιτύχετε. Εμείς σας δίνουμε κάποια στοιχεία για να κατανοήσετε πώς μπορείτε να επηρεάσετε το μέλλον και τι μπορείτε να κάνετε στα πλαίσια της πολιτικής σας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ja. Petra Ich bin jetzt mal Λοιπόν, Πραγματικά δεν καταλαβαίνω και είμαι πολύ ειλικρινής τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε. Κάπως έχω πάθει σύγχυση. So maybe I can answer with the um, um, one of the objectives of the study was really to provide... Σας απαντήσω. Προσπαθούμε να δώσουμε μια εικόνα του πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και να παρουσιάσουμε κάποια σενάρια και να απεικονίσουμε κατά κάποιο τρόπο το μέλλον για να δείτε ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις και με την πολιτική σας πώς μπορείτε να διαμορφώσετε κάποια πράγματα. Όλα αυτά δεδομένου ότι εσείς λαμβάνετε αποφάσεις. Και ανάλογα με τα αποφάσεις θα λάβετε πώς θα επηρεάσετε το μέλλον. Δεν θέλουμε να σας κάνουμε συστάσεις για το ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική σας ως Επιτροπή. So um, perhaps I can just add to that. So the idea of the να προσθέσω κάτι. Η ιδέα αυτών των διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων είναι να επιλεγούν κάποιες πολιτικές, κάποιες ιδέες. Δεν δίνουμε μία άμεση, αν θέλετε, συμβουλή. Κάποιες από τις ε, ιδέες που έχουμε βρίσκονται μέσα στην μελέτη αυτή και κατανοώντας καλύτερα ποιες είναι οι τέσσερις εναλλακτικές, καταλαβαίνετε εσείς σαν υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων πώς αυτό θα επηρεάσει το μέλλον. Μπορείτε να προβάλλετε κάποιες από αυτές τις λύσεις και να καταλάβετε καλύτερα, διαβάζοντας τη μελέτη μας, ποια θα είναι τα αποτελέσματα της επιλογής σας. Εσείς όμως μπορείτε να τα κατευθύνετε, να τα προσαρμόσετε και αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στο τι θα γίνει τα επόμενα 10-15 χρόνια. Ο κύριος Βέρ. Ήθελα να πω το εξή. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης και αυτό το οποίο αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε, πολιτική μας σε θέματα παιδείας. Βεβαίως ξέρουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία γεμάτη κινδύνους. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ποιο θα είναι το μέλλον όσον αφορά τις διάφορες εκπαιδευτικές πολιτικές, πολιτικές παιδείας γενικότερα. Σήμερα δεν υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των πολιτικών που ακολουθούνται σε θέματα εκπαίδευσης. Και οι δεξιά και οι σοσιαλιστές έχουν σχεδόν παρεμφερείς ιδέες για αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε αν αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν αυτές τις πολιτικές γνωρίζουν ποιες είναι οι προκλήσεις στις διάφορες κοινωνίες. Σήμερα ή αύριο. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε πάρα πολλές δυνατότητες που μας δίνονταν στον τομέα της εκπαίδευσης. Και πολλές φορές η άτυπη εκπαίδευση, η άτιμη παιδεία παίρνει όλο και περισσότερη σημασία. Όσοι έχουμε μικρά παιδιά, ξέρουμε πόσες πολλές πληροφορίες αποθηκεύουν από το ίντερνετ τα παιδιά. Ε, εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να προσπαθούμε ως πολιτικοί να λαμβάνουμε αποφάσεις με, το, με πιο πρωτοποριακό και ευφυή τρόπο. Έχουμε κάποια εκπαιδευτικά συστήματα που είναι καλά, υπάρχουν όμως άλλα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις. Χαίρομαι λοιπόν που μπορούν να μας βοηθήσουν τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα και μπορούν να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές σε τέτοιου θέματα να ακούσουμε ερωτήσεις και ενδεχομένως να μας δώσετε κάποιες πιο ουσιαστικέ πληροφορίες στις απαντήσεις σας. Ε, Herr Frankowski. Κυρία Φραγκόφσκι. Dziękuję za prezentację. Mam pytanie. Parlament Europejski, nasza komisja postulowała wielokrotnie wprowadzenie... Ευχαριστώ πολύ. Έχουν γίνει διάφορες ερωτήσεις εδώ στην Επιτροπή όσον αφορά την εκπαίδευση και τον ρόλο της ψηφιοποίησης. Θεωρούμε ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Το πιστεύετε σε αυτό? Η απάντηση είναι ναι αλλά είναι η προσωπική μου γνώμη. Δεν ε, το λάβαμε αυτό ε, υπόψη στο πλαίσιο της έρευνας μας, αλλά για να είμαι σύντομη, για μένα η απάντηση είναι ναι. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη σας. Έχω μία ερώτηση για την ίδια τη μελέτη γιατί πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα καλά τι θέλετε να μας δείξετε. Για να σιγουρευτώ λοιπόν. Στην αρχή παρουσιάσατε τα σενάρια προς τα που πηγαίνουμε και στη συνέχεια ποιες ήταν οι εναλλακτικέ πολιτικής. Αν τις εφαρμόσουμε λοιπόν και θα επαληθευτεί το σενάριο ή το αντίθετο. Γιατί εμείς εδώ σαν Επιτροπή θα έλεγα ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε την πολιτική και το αποτέλεσμα θα επηρεαστεί ανάλογα από το αν ε, διστάσει η Ευρώπη ή όχι. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν, ε, ε, το δικό μου σενάριο αυτό που προτιμώ είναι η ευθυγραμμισμένη Ευρώπη, επικεντρωμένη στους φοιτητές με ψηφιοποίηση κτλ αυτό που θέλετε λοιπόν να μας δείξετε είναι πώς εμείς ως Επιτροπής μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Um, so the idea of the scenarios is... Τα σενάρια αυτά ε, δεν θέλουν να σας... Ε, ε, στα παρουσιάσαμε για να έχετε ένα προτιμητέο σενάριο ή όχι, αλλά για να έχετε ένα σφαιρικό όραμα όσον αφορά την παιδεία αυτό που θέλαμε είναι λοιπόν να σας δείξουμε πολλές διαφορετικές πιθανότητες μελλοντικέ του πού μπορούμε να καταλήξουμε ανάλογα με τι, τι μπορεί να γίνει στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ήταν μια σύντομη παρουσίαση βέβαια και δεν μπορούμε να σας δώσουμε όλες τις ε, λεπτομέρειες, ό,τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τα σενάρια που σας παρουσιάσαμε εντάχει. Το θέμα είναι πώς συνδυάζοντας λοιπόν όλους αυτούς τους διαφορετικούς παράγοντες, οικονομία, εκπαίδευση κτλ. μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτά τα σενάρια. Και στη συνέχεια λοιπόν ανάλογα με την επιλογή πολιτικής έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Και εδώ μπορούμε να ερωτηθούμε, αυτό το σενάριο θα είναι επιτυχές, πώς μπορούμε να το επηρεάσουμε, τι χρηματοδότηση θα χρειαστούμε αν επιλέξουμε την διστακτική Ευρώπη ή την ευθυγραμμισμένη ανάλογα. Πώς μπορεί αυτή η πολιτική τελικά να είναι επιτυχήσα, άσχετα από το τι θα γίνει 15 χρόνια από σήμερα, αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά ποιες δράσεις μπορούμε λοιπόν να αναλάβουμε προκειμένου να κάνουμε τις πολιτικές μας επιτυχήσα και πώς μπορούν οι διαμορφωτές της πολιτικής να συνεργαστούν με άλλους παράγοντες σε άλλους τομείς και να επηρεάσουν έτσι τις αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα. Εμείς θέλαμε να σας δώσουμε κάποια μέσα για να προβληματιστείτε όσον αφορά τις επιλογές πολιτικής που έχετε σήμερα. Είναι υποθέσεις. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, την ψηφιακή εκμάθηση, για παράδειγμα, τι λέμε, τι νοούμε όταν λέμε ότι πρέπει να δώσουμε τους πόρους ε, έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, οι διδάσκοντες κτλ. Να σκεφτούμε λοιπόν πάνω σε όλα αυτά και να σκεφτούμε και τους κινδύνους. Εάν δεν εφαρμόσουμε αυτές τις επιλογές, ποιε θα είναι οι συνέπειες. Θα υπάρχουν λιγότεροι διδάσκοντες στις τάξεις. Θα είναι αυτό καλύτερο, γιατί η εκμάθηση θα είναι λοιπόν πιο φτηνή. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, αυτά τα εργαλεία σας δώσαμε. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι όσον αφορά το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μελέτη. Ή μπορείτε να επικεντρωθείτε περισσότερο στις επιλογές πολιτικής, δηλαδή κάθε ένα από αυτά τα σενάρια που σας παρουσιάσαμε και τα αναπτύσσουμε στην μελέτη να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα ποιες θα είναι οι συνέπειες της πολιτικής που θα υιοθετήσετε ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή μπορεί, μπορείτε να σκεφτείτε ποιο είναι το ε, αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε και στη συνέχεια να δώσετε προτεραιότητα ε, σε κάποιες πολιτικές επιλογές ή να επενδύσετε περισσότερο σε κάποιες άλλες. Η κυρία Φόξ. Um, despite the fact that you just... Παρά το γεγονός ότι εξηγήσατε λοιπόν την, τα σενάρια, δεν έχουμε και πολλά πράγματα για να βοηθηθούμε. Ακόμα και ο τίτλος νομίζω ότι θα έπρεπε ε, να παρουσιάσετε τα, να, τους τίτλους κάπως διαφορετικά. Νομίζω ότι δεν είναι καλό να μιλάμε για μια Ευρώπη που είναι σαν στρουθοκάμιλος. Είναι σαν να έχετε αποφασίσει εκ των προτέρων ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάρουμε. Βεβαίω η ευθυγραμμισμένη Ευρώπη, ναι, είναι μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη. Αν δείτε όμως αυτά που λέτε περί Ευρώπης ε, στρουθοκαμήλου, ότι ε, η οικονομία υποχωρεί, ότι το κάθε κράτο κλείνεται στον εαυτό του, υπάρχουν ε, κράτη-μέλη με ισχυρό κράτος που ξέρουν τι είναι καλύτερο για τους λαούς τους. Αυτή είναι μια θέση απομόνωσης, όμως εμείς θέλουμε μια δημοκρατία. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ουδέτερη η άποψή σας. Αυτά μας τα παρουσιάζετε πολύ ωραία, αλλά η γενική εικόνα είναι πολύ ζωφερή. Ε, ξεχάστε ότι είμαι Βρετανίδα και ότι υπάρχει το Brexit. Επικεντρωθείτε στην ερώτηση που έκανα. Νομίζω ότι το θέμα είναι αν θέλουμε να πάμε πολύ μακριά ή αν δεν έχουμε πάει αρκετά μακριά. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε κάνει την έρευνά μας αντελώς αμερόληπτα και ότι θέλαμε τα αποτελέσματά μας να είναι ουδέτερα. Είμαστε ανοιχτοί στην κριτική όσον αφορά και τον τίτλο των διαφορετικών σενάριων. Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα, αλλά οπωσδήποτε ε, προσπαθήσαμε να είμαστε ουδέτεροι. Άλλα ερωτήματα. Η κυρία Άντερσον, ναι. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Είναι σαφές ότι πολλά μέλη της Επιτροπής είναι εδώ και δεν μπορούν να κατανοήσουν ακριβώς τι θέλετε να μας πείτε με αυτήν την παρουσίαση. Και εμένα αυτό που συγκεκριμένα με εκνευρίζει είναι ότι υπάρχουν ε, τέσσερα σενάρια. Χρησιμοποιείτε δε κάποιες έννοιες τις οποίες εσείς κατανοείτε. Εγώ δεν ξέρω αν κατανοώ τι σημαίνει μια κατακαιρματισμένη Ευρώπη. Πρέπει να διαβάσω, να προσπαθήσω να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει αυξάνεται η ανεργία σε μια κατακαιρμένη Ευρώπη, μειώνεται ουσιαστικά το θετικό κομμάτι, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, και αυτή η οποία για μένα θα ήταν η έννοια της κατακαιρματισμένης Ευρώπης μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Βλέπουμε όμως ότι εσείς θεωρείτε συνώνυμα την Ευρώπη με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα όμως τα κράτη-μέλη δεν ε, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι όπως τα παρουσιάζεται, δηλαδή μειώνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται η ανεργία. Και αν κοιτάξω αυτούς τους τέτερις τίτλους σεναρίων, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείτε. Έχετε κάποια σημεία κλειδιά, μας λέτε πώς θα έπρεπε να είναι η κατάσταση εάν επιλέξουμε ένα από αυτά τα τέσσερα σενάρια. Γιατί όμως ε, με αυτό το σενάριο συμβαίνουν αυτά. Εγώ για μένα δεν είναι καθόλου σαφή οι επιπτώσεις. Πρόεδρος, να υπενθυμίσουμε και ποιος είναι ο τίτλος αυτής της μελέτης. Η μελέτη αυτή δεν αφορούσε το παρελθόν την κατάσταση στο παρελθόν. Σκοπός μας ήταν οι μελλοντικές προοπτικές. Αυτό ελπίζω να ήταν σαφές σε όλους. Να βασιστούμε δηλαδή σε κάποιες ε, πληροφορίες και δεδομένα του παρελθόντος, γιατί αυτό κάνατε για να μιλήσουμε για το μέλλον. Δεν ξέρω, μπορείτε να μου απαντήσετε και σε αυτό. So in, in terms of the uh, how we came to the four scenarios. Sorry. Um, so the, we started with actually Ξεκινήσαμε λοιπόν με 28 διαφορετικούς παράγοντες γύρω από την παιδεία και την οικονομία. Μελετήσαμε τα σχετικά άρθρα. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τους πιο σημαντικούς παράγοντες και προσπαθήσαμε λοιπόν να ε, κάνουμε μια ιεράρχηση αυτών των παραγόντων. Βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε και μια βεβαιότητα για κάποιους από αυτούς τους παράγοντες. Ε, εδώ μιλάμε για προβολές, προβλέψεις. Και προσπαθήσαμε να δούμε λοιπόν τη σχέση μεταξύ τους και να κάνουμε μία ανάλυση για το τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ε, εκμεταλλευτούμε την υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη. Προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε τα άκρα και να δούμε τα πιο ενδιαφέροντα σενάρια για να τεστάρουμε κάποιες πολιτικές επιλογές. Εάν δεν είχαμε συμπεριλάβει την κατακαιρματισμένη Ευρώπη, θα μας είχατε θέσει το ερώτημα γιατί δεν το κάναμε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες ε, στον εργασιακό χώρο, με τους νέους. Προσπαθήσαμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. Το σενάριο έχει μια ολόκληρη, είναι ένα ολόκληρο κείμενο, έχει και πολλά παραρτήματα. Προσπαθήσαμε να να συμπεριλάβουμε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που είναι σημαντικοί σε αυτό. Είναι πολύ σύντομος ο χρόνος για να μπορέσουμε να σας το παρουσιάσουμε, να σας παρουσιάσουμε τα σενάρια αυτά εκτενώς. Ε, είναι όμως αυτά τα σενάρια πραγματικά πολύ πιο εκτεταμένα, πάνε πολύ πιο μακριά. Προσπαθήσαμε να σας παρουσιάσουμε όμως τις πολιτικές και τους βασικότερους παράγοντες που εξετάσαμε. Να επικεντρωθούμε εκεί. Okay, thank you very much. Uh... Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πραγματικά δεν απαντήθηκε η ερώτησή μου. Εγώ ακόμα συνεχίζω να μην καταλαβαίνω τίποτα, να μην καταλαβαίνω τι είναι αυτή η κατακαιρματισμένη Ευρώπη, ποιες είναι οι επιπτώσεις, ποιες είναι οι συνέπειες. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Εγώ σας έδωσα ένα παράδειγμα. σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν μειώθηκε η ανεργία, ούτε σε όλες αυξήθηκε. Μπορείτε λιγάκι να με φωτίσετε. So, um, Όπως είπε και, λέει και ο τίτλος εδώ, ο τίτλος αυτού του σενάριου είναι «Και κατακαιρματισμένη Ευρώπη» όταν υπάρχει ε, κατακαιρματισμός δηλαδή, νομίζω ότι ε, η ερώτησή σας επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτό το σενάριο. Ε, θέλω να προσθέσω κάτι. Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τις πιο ευρείες επιλογές πολιτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν κάναμε συγκεκριμένη μελέτη χώρα με χώρα για να δούμε πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το κάθε σενάριο στις διαφορετικές χώρες μέλη. Α, όμως, όπως φαίνεται και από τα ίδια τα σενάρια, δεν λέμε ότι θα υπάρξει ή όχι αύξηση της ε, ε, απασχόλησης γενικά σε όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μιλάμε για μετακινήσεις μεταξύ των κρατών μελών, έχουμε λάβει υπόψη μας και την μετανάστευση, την εξέλιξη των τεχνολογιών και πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη με διαφορετικούς ρυθμούς σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Βεβαίως θα υπάρχουν λογικές διαφορές, τις έχουμε λάβει υπόψη μας. Ήταν πολύ δύσκολο ήδη να κάνουμε αυτή τη μελέτη σε επίπεδο ένωσης, και να έχουμε ένα επίπεδο βεβαιότητας. Προσπαθήσαμε λοιπόν ακριβώς να μην επικεντρωθούμε σε κάθε χώρα αλλά σε επίπεδο ένωσης, να βρούμε το μέσο όρο και έτσι γράψαμε, συντάξαμε αυτά τα σενάρια. Βεβαίως κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τα πάνε καλύτερα, κάποιες άλλες όχι. Ο κύριος Νίνας. Κοιτάξτε, Στη σελίδα 47 έχετε κάνει κάποιες ερωτήσεις. Στη σελίδα 61 βλέπετε κάποιες απαντήσεις για το θέμα της κατακαιρματισμένης Ευρώπης. 61, σελίδα 61. Η Julie Βόρτ ζητάει το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων που χρησιμοποιείτε τους εμπειρογνώμενες. Όλοι που έχουν πάει σε ένα πανεπιστήμιο διαπιστώνω ότι πρέπει να είστε πολύ ακριβείς και συγκεκριμένοι όταν ε, κάνετε μια τέτοια μελέτη και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ για να υπερασπιστείτε αυτό που κάνατε. Εγώ ήμουν επιχειρηματίας και καταλαβαίνω ότι αυτά τα σενάρια ουσιαστικά τα προτείνετε με την έννοια να εξουδετερώσετε κάποιες αρνητικές συνέπειες, κάποιους κινδύνους, κάποια πράγματα που δεν θέλουμε να συμβούν στο μέλλον. Μπορείτε να τα εφαρμόσετε ή να τα διανοηθείτε, να τα φανταστείτε σαν business σχέδια για την ε, ε, μελλοντική, αν θέλετε, εφαρμογή, υλοποίηση. Ιδιαίτερα για το θέμα της ψηφιοποίησης, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικά. Οι περισσότεροι εδώ εκτιμούν ιδιαίτερα αυτό που κάνατε. Ε, εννοείται ότι αυτό που κάνατε είναι ευρωπαϊκό. Εγώ νιώθω Ευρωπαία και χαίρομαι για την προβολή αυτών των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως την κάνετε. Έχω μία ερώτηση παρόλα αυτά. Είναι κάτι πολύ θετικό η ψηφιακή εξέλιξη. Απ' την άλλη υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι. Εμάς, ας πούμε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της γνώσης και της σωστής χρήσης αυτών των νέων τεχνολογιών στον ψηφιακό κόσμο. Τι ακριβώς έχετε να μας πείτε για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, για θέματα νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Πώς μπορούμε να καλύψουμε τα κενά που συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη θέση να μπορούν να καλύψουν το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους είτε αν παραδείγματο χάρη έχουν μόλις συνταξιοδοτηθεί αν βρίσκονται σε μια θέση απασχόληση η οποία τους επιτρέπει να έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο και θέλουν να συνεχίσουν να έχουν μια κατάρτιση, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, νέα προσόντα. Αυτό είτε στο πανεπιστήμιο είτε εκτός. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για την αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Apparently that was all going a bit wrong for the uh, translators. Είχαμε ένα θέμα με το μικρόφωνο. Ελπίζω εσείς να καταλάβατε την ερώτησή μου. Θέλω και εγώ να προσθέσω κάτι, λέει η Πρόεδρος. Όλοι θέλουν να έχουν συγκεκριμένες μελέτες για συγκεκριμένες περιπτώσεις και να μπούμε εις βάθος. Πριν λοιπόν επικρίνουμε τη μελέτη αυτή καθεαυτή, καλό θα ήταν να τη διαβάσουμε σε 15 λεπτά δεν μπορεί να παρουσιαστεί όλη αυτή η μελέτη, αλλά μπορείτε τώρα να μπείτε στην ουσία και να μπείτε σε κάποιες λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν τα μέλη. Uh, we on that. Δεν ασχοληθήκαμε στα πλαίσια αυτής της μελέτης με αυτό το θέμα. Αυτό όντως είναι κάτι το οποίο το έχουμε εξεχάσει, αλλά περισσότερο σε σχέση με την σχολική εκπαίδευση και όχι απαραίτητα με την ε, ε, μάθηση, την με φόρου ζωή. Πολύ καλά. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? sich mit der Studie ähm, auseinanderzusetzen und sollten daraus Fragen. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να διαβάσετε αυτή την ε, μελέτη που μας υποβλήθηκε για να έρχεται με τους υπεύθυνου σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη σας. Ευχαριστώ για τις διάφορες ε, εναλλακτικέ λύσεις, τα διάφορα σενάρια που μπορεί να αναπτυχθούν. Ευχαριστούμε επίσης για τις εξηγήσει που μας δώσατε. Αυτό που ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μας φωτίσετε για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη μελέτη που είναι η μελέτη που θα παρουσιάσει η κυρία Κλεμοντίν Ντομπεφ από το ΚΕΑ European Affairs και τον κύριο Ντονάτος Φούσιος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ποιοι ήταν οι στόχοι της μελέτης μας. Πρώτα-πρώτα θέλαμε να δημιουργήσουμε κάποια σενάρια τα οποία να είναι θετικά ή αρνητικά και επίσης να εντοπίσουμε τις διαφορετικές τάσεις εντός του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στην Ευρώπη, του CCS, και να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες ε, θα επηρεαστούν από αυτές τις τάσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο πολιτικής που έχει σχέση με ε, αυτούς τους ε, τομείς και στο τέλος να μπορέσουμε λοιπόν να διατυπώσουμε κάποιες συστάσεις για τους διαμορφωτές πολιτικής. Κάναμε μία ανάλυση των πραγμάτων όσα έχουν σήμερα ε, επίσης εξετάσαμε την σχετική βιβλιογραφία, συμβουλευτήκαμε ε, πολλές ενώσεις, δίκτυα, εμπλεκόμενα μέρη και επίσης το κάναμε αυτό για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο για τη μελέτη και τώρα ο συνάδελφός μου, ο κύριος Πόκιους, θα σας παρουσιάσει τα διαφορετικά σενάρια. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας πω εν συντομία πώς συντάξαμε αυτά τα σενάρια. Αναλύσαμε τη σχετική βιβλιογραφία το έκανε αυτό η συνάδελφος, ο Κλεμαντίν και άλλοι συνάδελφοι. Είδαμε λοιπόν τι υπάρχει στη βιβλιογραφία και μετά κάναμε δύο έρευνες, σε δύο φάσεις, μάλλον μία έρευνα σε δύο φάσεις. Επίσης, ένα, ε, απευθύναμε ερωτήσεις στον κλάδο, σε ενώσεις, σε εμπλεκόμενα μέρη. Είχαμε πάνω από 200 απαντήσεις. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος. Στο δεύτερο γύρο ε, με βάση αυτές τις απαντήσεις ε, κάναμε ένα εργαστήριο και με βάση τις απαντήσεις λοιπόν κάναμε, ε, καταρτήσαμε τα σχετικά σενάρια και τα αναπτύξαμε. Είχαμε ένα σύστημα μεμόρια για να πούμε ποιο ήταν το πιο πιθανό και ποιο το λιγότερο πιθανό σενάριο. Έχουμε λοιπόν κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Τα θετικά σενάρια, τα ενθαρρυντικά, είναι αυτά που επιθυμούμε περισσότερο και τα αρνητικά βεβαίως είναι αυτά που επιθυμούμε λιγότερο. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν τον τομέα της πολιτιστικής πολυμορφίας. Θα δείτε διάφορα σενάρια στις διαφάνειες, εγώ όμως θα σας παρουσιάσω κυρίως τα πιο πιθανά ή αυτά που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Όσον αφορά λοιπόν την πολιτιστική πολυμορφία, το πιο θετικό σενάριο είναι ότι ο τομέας λοιπόν ο δημιουργικός και πολιτισμικός, ο CCS, θα εκπροσωπεί διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και το ε, λιγότερο επιθυμητό είναι ότι ε, θα έχουμε πάρα πολλές πλατφόρμες και δεν θα μπορούμε πλέον να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Η αγορά εργασίας, το θετικό σενάριο είναι η διασυνορική κινητικότητα, κυρίως όσον αφορά τους επαγγελματίες αυτού του κλάδου. Θα αυξηθεί λοιπόν η κινητικότητα σε αυτό το σενάριο. Στο αρνητικό σενάριο όμως, οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό θα συνεχίσουν να εργάζονται με δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Όσον αφορά τώρα τις δεξιότητες και την εκπαίδευση, το θετικό σενάριο ο τομέας θα προαχθεί στην ε, κοινωνία και θα συμβαδίσει με τις ε, νέες, νεότερες τάσεις. Βρήκαμε όσον αφορά τα αρνητικά σενάρια μόνο ένα που δεν θεωρείται πολύ πιθανό από τους εμπειρογνώμενους που μπορεί όμως να επηρεάσει πάρα πολύ το μέλλον. Δηλαδή την έλλειψη χρηματοδότησης ε, και επαγγελματικών ευκαιριών που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερους επαγγελματίες σε αυτόν τον κλάδο. Η οικονομική βιωσιμότητα ε, ήταν κάτι που ε, συζήτησαν έντονα οι εμπειρογνώμονες τους οποίους συμβουλευθήκαμε. Το θετικό σενάριο είναι πολύ πιθανόν ε, ο τομέας CCS να παραμείνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην Ευρώπη, αλλά αυτό που μας ανησυχεί, αρνητικό σενάριο, είναι ότι ο τομέας θα εξακολουθήσει να έχει τεράστια έλλειψη χρηματοδότησης. Όσον αφορά το περιβάλλον, αηφορία. Θετικό σενάριο. Ο CCS θα αποτελέσει το έναυσμα για ατομική και κοινωνική αλλαγή. Όμως, αρνητικό σενάριο, τα μεγάλα δεδομένα και ε, το ψηφιακό αποτύπωμα θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία και αυτό θα είναι επιζήμιο για το περιβάλλον. Και τέλος, πολυμορφία και συμπεριληπτικότητα. Θετικό σενάριο. Ο CCS θα ενδυναμώσει την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Αλλά από την άλλη μεριά αρνητικό σενάριο θα έχουμε δημοκρατικές αλλαγές που θα μειώσουν την συμμετοχή στα CCS των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Η πρόσβαση λοιπόν στον πολιτιστικό τομέα θα παραμείνει πολύ δύσκολη, κυρίως στην περιφέρεια και τις αγροτικές περιοχές. Τελευταίος τομέας της ανάλυσής μας ήταν ο ρόλος των τεχνών και του πολιτισμού στις δημοκρατίες της Ευρώπης. Θετικό σενάριο, ο τομέα θα εξακολουθήσει να συμβάλλει στι κοινέ αξίες τη δημοκρατία, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ελευθερία τη έκφραση. Αρνητικό σενάριο θα υπάρξει αύξηση στην παραβίαση τη ε, ε, και μεγαλύτερη λογοκρισία έξι το δράσης, ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο δράση στα πλαίσια της εντολής σας. Αρχίζουμε με την πολιτιστική πολυμορφία. Πρόκειται για ένα κριτήριο στα πλαίσια της πολιτικής ανταγωνισμού. Θα πρέπει και στην εξελίξεις όλες και για την ε, ψηφιακή τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη να λάβουμε όλες αυτές τις πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές υπόψη. Σε θέματα ε, απασχόλησης στην αγορά εργασία θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους κανόνες της αγοράς ακόμη και για τις μη τυπικές μορφές εργασίας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα στάνταρ για τους αυτοαπασχολούμενους. Θα θέλαμε σε κάθε περίπτωση να έχουμε δυνατότητες συμπερίληψης των ε, τεχνών, των πολιτιστικών θεμάτων σε όλα τα ε, επίπεδα της εκπαίδευσης, σε όλα τα προγράμματα. Όπως ελέγχθη και στις προηγούμενες ερωτήσεις και απαντήτες, η πολιτική της ε, γνώσης προς όλους τους προθήσεις μπορεί να τους βοηθήσει να έχουν δημιουργικό και κριτικό πνεύμα. Όσον αφορά την βιωσιμότητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα οικονομικά κριτήρια, την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, θα πρέπει όλοι όσοι ε, συμμετέχουν στα, στην χρηματοδότηση να έχουν τη βιωσιμότητα και κατά νου να μπορούν στον τομέα τον πολιτιστικό και δημιουργικό να ακολουθούν φιλικές στο περιβάλλον περιοχές όσον αφορά τώρα την ε, διαφορετικότητα και την ε, συμπερίληψη θα πρέπει να υπάρχουν ερευνητικά έργα και μελέτες για το θέμα αυτό. Θα πρέπει πάντα να μπορεί καλής να ε, υποπτεύει και να μελετά το πώς ακριβώς ε, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλους τους μηχανισμούς οι οποίοι προωθούν την ισότητα των φύλων. Όλα αυτά θα μπορούν να γίνουν με την συλλογή δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρξουν Ε, σε όλες τις δημοκρατίες μας ή όλες οι διαδικασίες που θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλους να συμμετέχουν χωρίς αποκλεισμούς. Συστάσεις, προγράμματα, κλειδιά και πρωτοβουλίες, Creative Europe, Στρατηγική της Ευρώπης για θέματα πολιτιστικά, ώστε όλα τα δικαιώματα να εξασφαλίζονται. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια σαφής ε, γραμμή δράσης και τα απαραίτητα κονδύλια σε όλα τα επίπεδα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ευρώπης θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν στον τομέα μας και είναι θέματα στο πλαίσιο του Horizon Europe να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με την ε, νέα κοινότητα τεχνολογίας και καινοτομίας θα είναι έτοιμη το 2022 και θα πρέπει να γίνουν διάφορες προπαραβαστικές δράσεις σε επίπεδο CCC που θα συμπεριλαμβάνουν διάφορα κοινωνικού περιεχομένου νεοτηριστικά σχέδια. Ποια είναι τα κύρια μηνύματα η δημιουργικότητα είναι πρωταρχική σημασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που θα υπάρχουν στην ε, εργασία και στην ψηφιοποίηση των κοινωνιών. Ε, ένα υγιές CCC θα οδηγήσει σε δημοκρατικές, ανοιχτές και συμπεριληπτικές κοινωνίες στα πλαίσια των δημογραφικών αλλαγών. Το CCC Επίσης πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις τώρα. Madame Faron. Κυρία Φαγόν, ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα μελέτη που κάνατε. Όσον αφορά την διαφορετικότητα, καλό θα ήταν εάν ε, γίνεται να έχουμε και μεταφράσεις των εκθέσεών σας. Κρίμα, μόνο στα αγγλικά υπάρχουν. Ίσως υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στον ε, πίνακα με τα έξι σημεία. Όσον αφορά την ε, διάσταση της σημασίας των πολιτιστικών θεμάτων της Ευρώπης προς τα έξω καθώς και συμπερίληψη των, του οικονομικού σκέλους. Γίνεται στα πλαίσια της ΓΑΦ όλες αυτές οι συζητήσεις ε, για τα θέματα, αυτά τα θέματα της φορολόγησης και ακόμη και στο G7. Εκτός αν δεν κατάλαβα κάτι καλά στη μελέτη σας. Ίσως αυτό, αυτή η διάσταση λείπει. Εκτός εάν δεν το πρόσεξα σωστά εγώ. Θα σας απαντήσω αγγλικά. Στις συστάσεις, αυτό ίσως δεν το συμπεριλάβαμε, αλλά όταν μιλούμε για ίσες δυνατότητες για όλους και μιλούμε για την διεθνοποίηση και για τις τεχνολογίες στις, ε, στα κεφάλαια αυτά της έκθεσής μας το αναφέρουμε. Και όταν εμείς μιλούμε για τα πολιτιστικά κριτήρια και την διαφορετικότητα, αυτό εννοούμε. Στην σελίδα 46, θέματα της διεθνοποίησης. Σελίδα 46. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Καλύψατε το δύσκολο ερώτημα της ε, ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του τύπου και των μέσων, θέλω να κάνω ακόμα ένα βήμα. Πιο συγκεκριμένες συστάσεις, γιατί εδώ κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίζουμε δύο διαφορετικά φαινόμενα. Από τη μία προσπαθούμε να περιορίσουμε την ελευθερία έκφρασης σε πολλές χώρες, δεν θα τις κατονομάσω τώρα, ξέρετε τι εννοώ και την ίδια ώρα έχουμε τους λεγόμενους ε, ψεύτικες κατασκευασμένες ειδήσει. Φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, να περιορίσουμε, να αντιμετωπίσουμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας προς όλους αυτούς οι οποίοι δημιουργούν ψευδείς ειδήσει, κατασκευάζουν ε, ιστορίες χωρίς αντίκρισμα. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα αναφέρεται στις συγκεκριμένες συστάσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση, καθώς και τις δεξιότητες όσον αφορά το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Βεβαίως και το θέμα των ψευδών ειδήσεων αφορά άμεσα την απόκτηση δεξιοτήτων για να μπορέσει κάποιος να σκεφτεί με κριτικό πνεύμα και να μπορέσει να ξεχωρίσει τις αληθινές από τις ψευδείς ειδήσει. Η DigiConnect σίγουρα όσον αφορά το θέμα των έργων, των κινηματογραφικών έργων, αναφέρεται στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε τη σελίδα 18. Αφορά ακριβώς αυτό το θέμα. Και έχουμε και μία σύσταση που αναφέρεται σε μία πολύ στενή συνεργασία με τα αρμόδια όργανα για την ελευθερία και τη δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναφέρεται και σε διάφορα προγράμματα, τα οποία είναι προγράμματα για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων. Στηρίζουμε επίσης ε, την ενημέρωση μέσω πολιτισμικών διασυνδέσεων. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα πιο ε, σημαντικά σημεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Στακόφσκι. W imieniu grupy APP chciałbym podziękować za prezentację tych opracowań. Zapoznałem się z rekomendacjami tych badań. Ε, εμείς εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την σύσταση που κάνατε για την ε, πολυμορφία του πολιτισμού. Έχουμε το πρόγραμμα Creative Europe και θα ήθελα να σας κάνω την εξή ερώτηση. Στη μελέτη σας τίθεται και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Θεωρείται ότι είναι απειλή ή κάτι θετικό για την εξέλιξη ε, του πολιτισμού, κυρίως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμάς επίσης ως Ευρωβουλευτές μας ενδιαφέρει και το θέμα της χρηματοδότησης Έχουμε και εδώ διάφορα προγράμματα και έχουμε και τα διαρθρωτικά ταμεία ε, από που μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση για προγράμματα όπως το Creative Europe. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας και τις ερωτήσεις σας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι και απειλή και ευκαιρία. Γιατί μπορεί να είναι απειλή. Διότι κατά κάποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάκτηση περιεχομένου ή ε, να χρησιμοποιηθεί κατά της πολυμορφίας. Γιατί μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ε, συστήσει το ίδιο ακριβώς ε, περιεχόμενο, αρνητικό περιεχόμενο. Από την άλλη μεριά, μπορεί επίσης να βοηθήσει τους δημιουργούς να καταλάβουν καλύτερα τους χρήστες, πώς μπορούν να φτάσουν σε αυτούς πιο άμεσα και επίσης έχουμε και το θέμα της ε, κληρονομιάς, ε, της πολιτιστικής, το οποίο μπορεί να συμβάλλει. Το θέμα είναι να υπάρξει κατάρτιση, να βοηθήσουμε τον κλάδο να παραμείνει ανταγωνιστικός και να έχουμε συνεργασία μεταξύ ομάδων με διαφορετικές δεξιότητες. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη ε, θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή. Υπάρχουν όμως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τον τομέα αυτό. Όσον αφορά λοιπόν την ε, παιδεία, την κατάρτιση και την ε, καινοτομία θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα και επίσης χρηματοδότηση. Έχουμε το Creative Europe βεβαίως, αυτό το πρόγραμμα, αλλά και το Horizon Ευρώπη, στον δεύτερο πυλώνα που συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργικότητα. Έχουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο σε ολόκληρη την Ευρώπη για, να, για τη στήριξη των δημιουργικών τομέων. Και υπάρχουν όλο και περισσότερες περιφέρειες, λοιπόν, και όλο και περισσότεροι τομείς που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Το θέμα επίσης είναι να ε, έχουμε καλύτερο σύνδεσμο με τα προγράμματα COSME και το Erasmus ε, Συν. Ε, δεν το αναφέραμε εδώ πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν άλλες μελέτες που αναφέρουν ότι η συνεχής κινητικότητα, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνδέονται με το Erasmus Συν και επίσης η επαρκής χρηματοδότηση των προγραμμάτων, πολύ σημαντική, και να έχουμε αυτό το Ταμείο Εγγυήσεων για τον δημιουργικό τομέα. Και νέα επίσης εργαλεία χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνήθως δεν έχουν πρόσβαση στους παραδοσιακούς τρόπους χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν κάποιες που έχουν εφαρμοστεί, είχαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα και που στο μέλλον κυρίως ε, θα στηρίξουν ε, την δημιουργία. Κυρίως έχουμε το InvestEU. Θες να προσθέσεις κάτι. Ναι, ε, τα λέμε αυτά σε μία από την ε, σύστασή μας, ε, την τελευταία, όταν μιλάμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πώς μπορούμε να συνδέσουμε όλα αυτά με την κοινωνική καινοτομία και τις τοπικές κοινότητες. Uh, thank you. Yeah, thank you again for really interesting report. Um... Ευχαριστώ και πάλι για την ενδιαφέρουσα έκθεση αυτή. Εγώ έχω πενταετή θητεία σε αυτή την Επιτροπή και εδώ βλέπω την δουλειά της Επιτροπής, πράγματα τα οποία έχω πει, πρωτοβουλίες τις οποίες έχω λάβει. Αυτό λοιπόν που κάνετε εσείς είναι να αποδείξετε πόσο σημαντική δουλειά επιτελούμε εδώ στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Πόσο πιέζουμε για να ληφθούν σε επίπεδο Επιτροπής κάποιες πρωτοβουλίες. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα χρήσιμο έγγραφο αυτό, διότι μπορείτε να δείτε τι ακριβώς λέγεται, τι γίνεται και εκφράζεται και μία άποψη θετική για αυτό που κάνουμε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα το είχε πει η Επιτροπή και πολλοί κόσμοι ίσως δεν κατανοεί απόλυτα τι κάνουμε ε, εμείς ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που τα υπογραμμίζετε κάποια πράγματα από αυτά που κάνουμε εδώ. Ευχαριστώ, κυρία Παντένη. Αναφέρομαι στη σελίδα 78. Γίνεται λόγος για το γεγονό ότι στον δημιουργικό τομέα των αυτοπασχολούμενων, των freelance που εργάζονται βάσει προγραμμάτων. Αυτό ε, που, η περιγραφή που κάνετε είναι πάρα πολύ πραγματιστική, τουλάχιστον δηλαδή, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, εγώ έχω εργαστεί ως freelance σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και η ερώτησή μου είναι μπορείτε να κάνετε κάτι για να ενθαρρύνετε τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν άτομα ως freelance. Βεβαίως, στις ε, μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι ίσως ε, ε, τα πράγματα διαφορετικά. Στις μικρότερες είναι πιο ανθρώπινα είναι πιο προσωπικά. Διότι αν κάποιος δεν έχει ασφάλεια για το τι θα κάνει όταν τελειώσει το πρόγραμμα και αν δεν υπάρχει ένα επόμενο, δεν είναι ίσως τόσο πολύ θετικός και δεν είναι πάρα πολύ δημιουργικός. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή λέτε ότι είναι ε, καλύτερο να είναι κανείς αυτοαπασχολούμενος freelance σε μεγάλες επιχειρήσεις, να μου το εξηγήσετε κάπως περισσότερο. Εξαιρετική όμως η εκθέση σας, ευχαριστώ. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν έχουμε μεσαίου μεγέθους πολλές επιχειρήσεις εδώ. Έχουμε μικρομεσαίες και μεγάλες, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε τα παραδείγματα. Και υπάρχουν ορισμένες ακόμη και μονοπρόσωπες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να επιτύχουν παρά μόνο εάν διάφορα άτομα ενώσουν τις δυνάμεις τους. Και υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία εργάζονται ε, σε στεγανά, μόνα τους. Εάν μπορούσαν όλοι λοιπόν να συνεργαστούν και να εποφελούνται μένα από τους δε, αν μπορούσαν να δημιουργήσουν νέους τρόπους, δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καλύτερα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του τομέα στον οποίο υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις και αν κάποιος είναι ε, δημιουργικός μπορεί ακόμη και σε επίπεδο μικρής επιχείρησης να κάνει κάτι που να βοηθήσει να αναπτυχθεί πολύ η επιχείρηση. Ευχαριστώ. Κύριε Νίκλας, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Εύκολα σας παρακολούθησα. Έχω μια ερώτηση για την ε, μελέτη σας σε σχέση με την παρουσίαση που κάνατε τσέκαρα αυτά τα δύο και τα σενάρια που παρουσιάσατε και τις διάφορες κατηγορίες δεν τις βρίσκω μέσα στη μελέτη σας. Μπορείτε λοιπόν να μου πείτε πώς από αυτή την περιληπτική παρουσίαση μπορούμε να βρούμε περισσότερα στοιχεία πιο λεπτομερή μέσα στη μελέτη σας. Um, speaker before me. Um, Επίσης, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι πριν, εξετάσατε το ότι αν έχει κανείς λιγότερους πόρους τον εμποδίζει από το να είναι πιο δημιουργικός και εδώ τι ρόλο έχουν να παίξουν οι freelance για κάποια επιχείρηση. Το πρώτο θέμα σας. Σελίδα 60. Έχετε τα σενάρια σε σχέση με τον ε, εργασιακό τομέα, τον οικονομικό. Έχετε τη ε, θετική προσέγγιση, την αρνητική. Και βεβαίως όλα αυτά με διάφορους δείκτες ε, πιθανοτήτων και ποσοστά. Στην παρουσίαση σε ορισμένες περιπτώσεις εστιάσαμε σε λιγότερα στοιχεία, διότι θελήσαμε να είναι σύντομη αυτή η παρουσίαση. Αλλά στη σελίδα 60 βλέπετε όλα τα σενάρια που ακολουθούνται και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, στη σελίδα 8 που έχετε τη συνοπτική παρουσίαση έχετε τα διάφορα σενάρια ανακατηγορία. Δεν υπάρχει το θέμα της ε, πολιτιστικής διαφορετικότητας, αλλά υπάρχει το θέμα της ελεύθερης έκφρασης στις διάφορες δημοκρατικές χώρες και κυρίως Προσπαθήσαμε να είμαστε πιο συνοπτικοί στην παρουσίαση, γι' αυτό ίσως δεν βρίσκεται την, ε, τον παραλληλισμό. Σύντομα, για να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά σας. Το να είναι κανείς ε, φτωχός, ε, να έχει λιγότερα κονδύλια σημαίνει ότι είναι και πιο δημιουργικός. Δεν βρήκαμε απόλυτη διασύνδεση μεταξύ αυτών των δύο. Αλλά αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ένας κατακαιρματισμένος τομέας είναι να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και υπάρχουν δημιουργικοί άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές απασχολούνται και σε χιλιάδες άλλα πράγματα. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι η δημιουργική εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ε, επαγγελματικά προσόντα, αλλά να έχουν και κάποιες δεξιότητες σε θέματα ε, διοικητικής διαχείρισης της δουλειά την οποία κάνουν, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν περισσότερο με το δημιουργικό κομμάτι της εργασίας τους. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Προ το παρόν σας ευχαριστούμε πολύ για τι παρουσιάσει σας και θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο σε αυτό το στάδιο. Yes. Uh, thank you. No particular comments just to Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε ιδιαίτερα σχόλια. Θέλαμε απλώ να πούμε ότι και για μας η έκθεση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ήταν πολύ ενδιαφέρον που μας δείξατε πώς όλα αυτά σχετίζονται με το πολιτιστικό θεματολόγιο της Ευρώπης για το 2020 και έχουμε και ένα σχέδιο εργασιών ε, για τον πολιτισμό στην Ευρώπη 2020 και όλα αυτά βεβαίως θα τα εφαρμόσουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, για το ότι ήρθατε εδώ σήμερα. Και τώρα θα κάνουμε μισή ώρα διάλειμμα, γιατί ο Επίτροπος κύριος Ναύρατσικς δεν θα έρθει εδώ πριν από τις 5. Αυτό είχαμε αποφασίσει αρχικά. Μπορείτε λοιπόν να πάτε για έναν καφέ. Du wolltest mit mir über Doris Pack reden. Ja, also müssen wir nicht jetzt machen, aber wir müssen ja, auf jeden Fall irgendwie... Ähm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 Ladies and Αγαπητοί συνάδελφοι, για όλους όσους έχουν επανέλθει, ξέρω δεν είναι εύκολο πάντα όταν διακόψουμε το να σας ξαναφέρουμε μέσα στην αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να περιμένει ο Επίτροπος περαιτέρω. Καλώς ορίσατε, κύριε Επίτροπε, κύριε Ναύρατσιτς. Είσαστε στην τελική φάση της θητείας σας σαν Επίτροπος και είναι μεγάλη χαρά για μας που θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας να ακούσουμε τι έχει εκπληρωθεί, ποια είναι τα υπόλοιπα που θα κάνετε και πώς βλέπετε το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε μαζί μας για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκλογή σας. μια πολύ σημαντική ανανέωση του ευρωπαϊκού πνεύματος και της ευρωπαϊκής δημοκρατικής διαδικασίας. Συγχαρητήρια λοιπόν. Θα ξεκινήσω με μια λίγο πιο μεγάλη εισαγωγική παρουσίαση, περισσότερο από ό,τι συνήθως. Πλησιάζουμε το τέλος της θητείας μας, θητεία αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μια σύνοψη, να παρουσιάσουμε τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα αυτής της περίοδου. Ίσως λοιπόν ε, πάρω το λόγο για λίγο περισσότερα λεπτά από ό,τι συνήθως. Το να είναι κανείς υπεύθυνο για τους νέους, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, είναι κάτι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πραγματικά η συνεργασία μαζί τας ήταν εξαιρετική. Το να μπορέσει κανείς να επενδύσει τους νέους, στη νεολαία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε αυτά αποτελέσματα. Ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, οι νέοι και ο αθλητισμός παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας Ευρώπης που ξεπερνάει τον εαυτό της και που βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. Ουσιαστικά μπορούμε και δημιουργούμε μια νέα κοινωνία. Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι οι κοινέ μας αξίες, ο πολιτισμός μας και μπορούμε να ενισχύσουμε και την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή παιδεία το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σύστημα μέχρι το 2025 θα κάνει πολύ σημαντικά βήματα για όλους τους νέους, για όλους τους σπουδαστές που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε σε νέα επίπεδα ανταλλαγών. Ανοίγουμε νέες ευκαιρίες ήδη από τώρα. Σε ένα χρόνο μάλλον ένα χρόνο μετά το 2017, όταν για πρώτη φορά οι ηγέτες της Ευρώπης πήραν αυτή την απόφαση, περάσαμε στην αμοιβαία αναγνώριση των ε, πτυχίων, την αναγνώριση των ε, προσόντων στον ψηφιακό τομέα, και την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης τη διδασκαλία. Τα κράτη-μέλη επίσης έχουν δεσμευθεί έτσι ώστε να προωθήσουν την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών στο τέλος ε, της ε, φάσης της ανώτερης εκπαίδευσής τους. Θα πρέπει πολύ νωρίς να ξεκινάνε αυτές οι ε, εκπαιδευτικές διαργασίες. Όσο νωρίτερο, τόσο καλύτερο. Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές δεξιότητες και προσόντα, έτσι ώστε να μπορούν οι νέοι μας να σκέφτονται με κριτικό πνεύμα, να προσαρμόζονται στην ε, νέα τεχνολογία και να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους ε, νέους από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως υπάρχουν και αντικρώμενα συμφέροντα και πολλές φορές κάποιοι φοβούνται και δεν βλέπουν όλες αυτές τις εξελίξεις σαν αλλαγές. Και μάλλον θέλουν να συρρυκνώσουν τις δυνατότητες, να περιορίσουν την επικοινωνία και όχι να ανοιχτούν προς τα έξω. Εγώ πολύ νωρίς, το Μάρτιο του 2015, υπέγραψα την ε, Συμφωνία του Παρισιού με όλους τους Υπουργούς Παιδείας με σκοπό να στηρίξουμε τις κοινέ μας ευρωπαϊκές αξίες, να δημιουργήσουμε νέο περιβάλλον για τους Ευρωπαίους βάση του Erasmus Plus και περισσότερων ανταλλαγών. Επίσης κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα όσον αφορά την ενίσχυση των κοινοτήτων των νέων. Δίνουμε νέες ευκαιρίες πριν από δύο μήνες ανακοίνωσα το, το 17ο συνέδριο με σκοπό να προωθήσουμε αυτά τα προγράμματα που στηρίζουν και προωθούν την ευρωπαϊκή κοινότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Καλύτερες ευκαιρίες και δυνατότητες για τους φοιτητές από όλες τις κοινωνικές ομάδες να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σαν Ευρώπη, σαν ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να ξεκινήσουμε τη νέα πειραματική φάση. Βεβαίως όλα αυτά στηρίζονται από ένα ενισχυμένο πρόγραμμα Εράσμους. Γιορτάσαμε το 17 το 30 έτος από το ξεκίνημα αυτού του ε, προγράμματος Εράσμους με εκατομμύρια Ευρωπαίους φοιτητές και σπουδαστές οι οποίοι έχουν υποφεληθεί και χρησιμοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Θέλουμε να το κάνουμε πιο εύκολο στην πρόσβασή του για όλους. Πρόκειται για ένα συμβολικό πρόγραμμα. Μπορούμε να το βελτιώσουμε και συμφωνώ απολύτως με τη φιλοδοξία σας να το κάνουμε προσβάσιμο σε περισσότερους νέους της Ευρώπης, να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες, να μάθουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό με περισσότερες ε, πιο ευέλικτες δυνατότητες. Και βεβαίως να ε, βοηθήσουμε μικρούς φορείς να επωφεληθούν. Πιο ανοιχτός τρόπος να ανακαλύψει κάποιος την Ευρώπη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επιτρέπει σε παιδιά 18 ετών, 1500 ε, παιδιά από όλη την Ευρώπη, να επωφεληθούν από μία διαμονή και σπουδέ στο εξωτερικό, να γνωρίσουν τι είναι η πολυμορφία, η πολιτισμική και οι κοινέ μας αξίες. Όσον αφορά τη διδασκαλία το Discover EU είναι κάτι που θα ενσωματωθεί και θα αποτελέσει τμήμα του Erasmus Plus στο μέλλον. Υπάρχει πραγματική δυνατότητα να κερδίσουν οι νέοι Ευρωπαίοι εμπειρία και να επωφεληθούν από περισσότερες ε, δυνατότητες, ε, ευκαιρίες διαμονής και σπουδών στο εξωτερικό. Και αυτό όχι μόνο μέσω του Εράσμους, αλλά και μέσω των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους. Νέες ευκαιρίες για την νεολαία να περάσει μέσα από αυτές τις ε, εμπειρίες στο εξωτερικό, να αυξήσει τις δεξιότητές της και να επωφεληθεί 157.000 νέοι έχουν επωφεληθεί. Πάνω από 20.000 έχουν δραστηριοποιηθεί, δημιουργώντας περισσότερη κοινωνική συνοχή. Θέλουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης να ενισχύσουμε τις δυνατότητες και τις δράσεις μετά το 2020, δίνοντας πολύ περισσότερες ευκαιρίες ακόμα και στην εθελοντική δράση. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δίνει δυνατότητες στους νέους να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως ε, συμβαδίζει με τις γενικότερες πολιτικές και στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υλοποιηθούν από φέτος. Ένας κεντρικός σκοπός είναι να ενισχύσουμε το διάλογό μας με τις νέους, περισσότερες προσπάθειες να έχουμε πρόσβαση σε όλους, ιδιαίτερα όλους αυτούς που δεν ανήκουν σε οργανώσεις νεολαίας, όλοι αυτοί που ζουν περιθωριοποιημένοι ή απομονωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό για τους νέους να γίνουν γνωστές οι δυνατότητες προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εισακουστούν οι φωνές τους και τα σχέδιά τους. Από το 14 μέχρι το 19 έχουμε έτσι προσεγγίσει πολλές χιλιάδες νέους. Αυτό είναι σημαντικό μέρος της εργασίας μου και ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θέλει να αρχίσει διάλογο και έχει διάλογο με τους νέους. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι δραστηριότητες που βοήθησαν και τόσους πολλούς νέους να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές το Μάιο. Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσω τώρα σε θέματα αθλητισμού. Το να ε, προωθήσουμε την ε, υγιεινό τρόπο ζωής και την άθληση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και με τους ε, συναδέλφους από την Γεωργία και την ε, Υγεία, τους συναδέλφους επιτρόπους Κάναμε ένα πρόγραμμα το 2017 που να συμπεριλαμβάνει αυτά τα θέματα. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου επίσης θέσαμε σε κίνηση την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Ε, φέτος σε λίγες μέρες θα αρχίσει η νέα εβδομάδα του έτους στην ε, Φινλανδία και βοηθούμε τους νέους να είναι πιο ενεργοί και να ασχολούνται με την γυμναστική και τον αθλητισμό διότι δεν είναι μόνο θέμα ευημερία. Είναι ένα, μια σημαντική δραστηριότητα η οποία δεν ε, υπολογίζει τις ε, κοινωνικές, τους κοινωνικούς φραγμούς και τα εμπόδια, βοηθάει περισσότερο τους νέους και βοηθάει και την ε, κοινωνική συμπερίληψη. Το μέλλον των προγραμμάτων Erasmus Plus θα προστε προσφέρει και νέα κονδύλια ώστε να μπορέσουμε και από τις ρίζες να προωθήσουμε πιο υγιεινή ζωή. Η... Τα θέματα τα πολιτιστικά είναι πάλι μία από τις προτεραιότητες ε, της ε, ατζέντα της Νέας Επιτροπής. Το 2017 η Αρχή Κρατών και Κυλήσεων είπαν πόσο σημαντικό είναι τα θέματα τα πολιτιστικά και υποστηρίζουν τα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και δημιουργικότητα. Για το 2019-2024 ζητείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να προσφέρουν περισσότερα κονδύλια σε θέματα πολιτιστικά. Είμαι υπερήφανο διότι κάτι τέτοιο έγινε χάρη και στι δικέ μου προσπάθειε. Το 2018, με την νέα ατζέντα για πολιτιστικά θέματα, δώσαμε νέα όθηση σε μια, στη νέα πολιτιστική ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε προωθήσει νέες ε, πρωτοβουλίες με θέματα πολιτιστικά για νέους κανόνες για τους δημιουργούς, σε θέματα καινοτομίας, σε θέματα ψηφιοποίησης. Κάτι άλλο το οποίο έχουμε κάνει εγκρασίως είναι να προσφέρουμε το νέο Ινστιτούτο για την ε, τεχνολογία και την έρευνα που τα τελευταία δέκα χρόνια έχει γίνει το, ε, αποτελέσει το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης την ε, λειτουργία για ένα νέο δικτύο το 2021. Είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεισφέρει ε, στην δημιουργία ε, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και θα οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας. Το 2018 περισσότερο από 6,2 εκατομμύρια άτομα συμμετείχαν σε ε, περισσότερους από 1.000 πολιτιστικές εκδηλώσεις, 11.000 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συγγνώμη, στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, νομίζω ότι υπογραμμίζεται και ο ρόλος του πολιτισμού ε, στην, ε, και της πολιτιστικής κληρονομιάς για όλους εκτός από την ε, προσφορά της κουλτούρας στις κοινωνίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνουμε και για μας και για τους νέους για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον αύριο το Ευρωπαϊκό της Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι κάτι το οποίο ε, γίνεται κάθε χρόνο. Προτε, προτάθηκαν περισσότερο από 60 δράσεις του τέλους του 2018 και ακόμη περισσότερες τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω τελειώνοντας για το πρόγραμμα Creative Europe. Με πολλές εκατοντάδες οργανώσεις οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα. Εκτιμούμε ότι έτσι έχουμε προσεγγίσει περισσότερα από 77 εκατομμύρια άτομα με όλες τις πρωτοβουλίες του Creative Europe. Και νομίζω ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση και πρέπει να υπάρχει και μακροπρόθεσμα στον κοινοτικό προϋπολογισμό για να συνεχιστούν τέτοιες δραστηριότητες. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι διότι πάντα με υποστηρίζετε στα πλαίσια της πολιτικής μου με ενθουσιασμό. Ήταν η αποφασιστική συνεισφορά σας για να μπορέσει να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκά τους πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και άλλες πρωτοβουλίες. Πιστεύετε στους νέους και αυτό είναι κάτι το οποίο σας όθησε και να κάνετε το πρόγραμμα αλλαγής για τους νέους ακόμη και σε οικονομικά δύσκολους κερνούς. Πιστεύω ότι ε, μπορώ να πω ότι πάρα πολλές από τις πρωτοβουλίες μας τις έχετε ενστερνιστεί. Όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να, μπορέσουν, ε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προγράμματά μας. Έχετε καταλάβει πώς εμείς εφαρμόζουμε τα προγράμματά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας. Εσείς αρχίζει μια νέα θητεία, η δική μου τελειώνει. Τις επόμενες εβδομάδες θα ε, περάσουμε σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων για προγράμματα νέας γενιάς. Και νομίζω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να προωθηθούν όλα τα προγράμματα εκπαίδευση, όλα τα προγράμματα ε, που αφορούν τον ε, αθλητικό τομέα και ό,τι μπορεί να οδηγήσει στην ευημερία των νέων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα σας ευχαριστώ για την ε, εξαιρετική συνεργασία που είμαι. Εύχομαι το ίδιο να συμβεί και με τον διάδοχό μου στη θέση του Επιτρόπου για θέματα πολιτιστικά. Ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Ερωτήσεις. Α, έχουμε ήδη ένα κατάλογο. Ξεκινάμε με την Μιχαέλα Ζόντροβα που είναι και η συγγήτρια. Ε, και συντονίστρια, συγγνώμη. Jeho zhrnutí uplynulých pěti let. Vy jste sám e, velmi dobře vyjmenoval to, co e, vnímáte jako úspěšný. Επίτροπε, αναφερθήκατε στις επιτυχίες, στις πρωτοβουλίες που πέτυχαν Γιορτάσαμε τα 30 χρόνια του Εράσμους πριν από λίγα χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο δείξαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία του προγράμματος αυτού που έχει σταθεροποιηθεί, έχει επιβληθεί, προτείνουμε να διπλασιαστεί ο προπολογισμό του. Και αυτό δείχνει ότι η συνεργασία της Επιτροπής μας με τις υπηρεσίες της Επιτροπής σίγουρα θα έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Και ουσιαστικά αυτά που λέτε μας οδηγούν στο να ζητήσουμε ενδεχομένως και τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος. Υπάρχει ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης, αυτό είναι δεδομένο. Άλλο πρόγραμμα, το Creative Europe, που έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στο έτος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, την οποία γιορτάσαμε. Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στο Creative Europe συνεχίζουν να αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα και μπορώ να σας δώσω και πάρα πολλά παραδείγματα σχολείων που έχουν επωφεληθεί από αυτά τα προγράμματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί στηρίζετε επίσης και την ε, επιχειρηματικότητα και κυρίως τον τομέα που αναφέρατε και στην ομιλία σας του αθλητισμού και τον ευεργετικό ρόλο που παίζει ο αθλητισμός στους νέους. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω για την στήριξη στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Κάτι που πραγματικά στηρίξατε από την αρχή. Ακούσατε τα σχόλιά μας, τα ενστερνιστήκατε ακούσατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη αυτού του εγχειρήματο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι προσδοκίες μας έχουν ε, εισακουστεί και για τη νέα περίοδο βεβαίως έχουμε πολύ πολλές ε, προσδοκίες και ελπίδες. Μπορείτε να μας πείτε Ποιο είναι αυτό που θα θέλατε να στηρίξετε για το μέλλον, τι είναι αυτό το οποίο κατά την άποψή σας είναι τόσο επιτυχημένο που πρέπει να συνεχιστεί. Um, my legacy to be continued το πιο σημαντικό μέρος το οποίο θα ήθελα να αφήσω για να το ολοκληρώσει ο διευθυντικός μου είναι τα προγράμματα για τα θέματα τα εκπαιδευτικά. Πρόκειται για τις ίδιες αρχές. Είδαμε πώς είναι οι προσανατολισμοί για το μέλλον, αλλά θα πρέπει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να γίνουν μια πραγματικότητα. Τώρα αρχίζουμε. Πρέπει να πω ότι θα πάω σε ένα από τα πρώτα σεμινάρια, ένα πραγματικό σεμινάριο, ένα workshop που θα οργανωθεί ε, από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σε, θέματα τεχνών, αλλά θα πρέπει όλες αυτές οι συμμαχίες που έχουν δημιουργηθεί να γίνουν πραγματικά πανεπιστήμια. Και θα πρέπει βεβαίως να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, όπως λέει και η Φινλανδική Προεδρία, της διαβίου μας μάθησης, Πρώτη καλή ευκαιρία θα δοθεί στις 8 Νοεμβρίου όταν θα γίνει ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας και βεβαίως χρειάζονται και τη δική σας υποστήριξη και τις δικές σας υποδείξεις και προτάσεις. Αν έπρεπε λοιπόν να επιλέξω ένα τομέα, θα επέλεγα τον τομέα της εκπαίδευσης, της παιδείας, διότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Αποτελεί την βάση της στενότερης ενεργασίας μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ διαφόρων ε, κοινοτήτων και μπορεί να επηρεάσει και την πολιτιστική ε, πολιτική, την πολιτική για την νεολαία. Ε, Ευχαριστώ κυρία Κάμερβελ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνεται πολύ συγκεκριμένα ότι παρόλες τις έντονες πολλές φορές αντιμαχίες και ανταλλαγές απόψεων που είχαμε εδώ, πετύχαμε κάποια πράγματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Μιλήσατε για το σχέδιο του Κοινοβουλίου για το έτος ε, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης Ξέρετε ότι κατά κάποιο τρόπο ανησυχούμε να μην επιβραδυνθούν αυτά τα προγράμματα ακριβώς επειδή κάποια κράτη-μέλη θα επωφεληθούν από αυτήν την μεταβατική περίοδο για να εγκαταλείψουν αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να στηρίξουμε αυτούς τους κοινούς μας ε, στόχους και ελπίζω με τον διάδοχό σας ή με την διάδοχό σας από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν στους τομείς αυτούς έτσι ώστε με το θέμα αυτό αν θέλετε, δεν θα γίνει θέμα αντιπαράθεσης αρμοδιοτήτων από τη μία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την άλλη των κρατών μελών. Χρηματοδότηση του Erasmus Plus. Ναι, η Επιτροπή ζήτησε διπλασιασμό των κονδυλίων. Εγώ θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν εσείς και ο η διάδοχός σας στηρίζατε την πρότασή μας να τριπλασιαστούν τα κονδύλια και να πείσετε τα κράτη-μέλη αυτά που διαφωνούν ότι αυτό είναι ε, η πρόταση η οποία πρέπει να περάσει. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, η πρωτοβουλία να προωθήσουμε και να στηρίξουμε την αριστεία, όλα αυτά τα οποία στηρίζουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται πολύ επεξεργασία ακόμα βεβαίως. Είμαστε σε μια φάση σχεδιασμού ακόμα. Αυτά τα τρία όμως σχέδια πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένα. Πρέπει να αξιολογήσουμε τα πιλωτικά προγράμματα, αυτό είναι σαφές. Και Τα τρία αυτά επαναλαμβάνω σωστά προγράμματα, ισχυρά προγράμματα να τα δούμε να υλοποιούνται. Και μια προσωπική παρατήρηση, κύριε Επίτροπε. Τα πέντε χρόνια αυτά που πέρασαν, όντως είχαμε έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, αλλά κάθε φορά βρήκαμε τρόπο να συνεργαστούμε επικοδομητικά και θυμάμαι ότι σαν πρόεδρος είχα πολλές συζητήσεις μαζί σας και θέλω σήμερα από την καινούργια μου θέση να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω γιατί πάντα βρήκαμε έναν λογικό και επικοδομητικό τρόπο να συνεργαστούμε παρά όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ο Επίτροπος. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, χάρηκα τόσο τις α, αντιπαραθέσεις μας όσο και τις συμφωνίες μας στο παρελθόν. Ε, είχαμε μια θυελώδη αρχή, θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά αναπτύξαμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία με όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα περήφανος ε, για αυτόν τον συνεχή διάλογο και την επικοδομητική μας συνεργασία. Όσον αφορά τον ε, Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε Υπάρχει η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, ε, υπάρχει αυτό το θέμα βέβαια, και ακόμα και στο πρόγραμμα έρασμου, το θέμα το σύστημα των μορίων και της αναγνώρισης δεν είναι πάντα πολύ εύκολο. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε λίγο-λίγο όλες αυτές τις δυσκολίες. Και όσον αφορά το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, αυτό μπορεί να δώσει μια μεγάλη όθηση στην ανώτατη παιδεία. τα αμοιβαία ωφέλη της συνεργασίας είναι πολύ σημαντικά και ε, τα κράτη-μέλη ε, θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις διαφορές και τις υποψίες τους. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση από τις επιχειρήσεις, από την, τον οικονομικό τομέα, διότι η εκπαίδευση σήμερα στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένη. Υπάρχουν 50 διαφορετικά συστήματα παιδείας στην Ευρώπη, 16 στη Γερμανία, πολλά στην Ισπανία, όπου η πολιτική, η εκπαιδευτική καθορίζεται σε επίπεδο περιφερειών. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες καλές λύσεις για να μπορέσουμε να συντονίσουμε και να εναρμονίσουμε ε, την προσέγγιση μας, να εναρμονίσουμε αυτά τα διαφορετικά συστήματα. Είχαμε λοιπόν βεβαίως τους τριμερείς, έχουμε τους τριμερείς διαλόγους και τις χρηματοδοτικές λύσεις. Βλέπουμε, προσβλέπουμε προς το μέλλον, αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε περισσότερα προγράμματα και ότι εγώ και η ε, διαδοχή μου θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτά τα προγράμματα. Αυτό που είναι ξεκάθαρο για μένα και την υπηρεσία μου είναι ότι χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα και το Erasmus και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Creative Europe, ούτως ώστε να ε, έχουμε μια πιο συμπεριληπτική παιδεία και κοινωνία και να μπορέσουν όλοι να λάβουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα. Ελπίζω λοιπόν ότι οι διαδοχή μου θα συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο. Όπως είπα, είχαμε μια κάπως δύσκολη αρχή, αλλά στη συνέχεια συνεχίσαμε με αγαστή σύμπνοια. Η κυρία Φαγάνς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτόν τον απολογισμό, πολύτιμο για μας, τους νέους βουλευτές είμαι και εγώ καινούρια εδώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την διάσταση του πολιτισμού. Είναι και παράγον συνοχής, είναι το τσιμέντο κατά κάποιον τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σε, στην σημερινή περίοδο με το Brexit. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι για μένα σημαντικό. Υπάρχουν πολλά βραβεία που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, το βραβείο Λούξου για παράδειγμα, που είναι επιβράβευση για ποιοτικά έργα. Όμως τα έργα αυτά δεν έχουν την ανάλογη προβολή αυτή που θα άξιζαν εντός της Ένωσης. Πιστεύετε ότι υπάρχουν μέσα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καλλιτέχνε τη, ο πολιτισμό τη να γίνει ένα πραγματικό σήμα ποιότητα, το οποίο να μπορούμε να διαδώσουμε και να μοιραστούμε περισσότερο. Επίση, όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι πολύ σημαντική η πολιτιστική κληρονομιά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το κοινό μας παρελθόν, που είναι και πηγή περηφάνειας. Για μένα υπάρχει εδώ κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε περισσότερο τον τομέα αυτό. Και θα ήθελα να μάθω ποιες ε, φιλοδοξίες θα μπορούσαμε να έχουμε επί του θέματος. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά για την μεγαλύτερη συμμετοχή και το κοινό πρόγραμμα ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης και το Creative Europe. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Ένα μέρος της Creative Europe έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλες λοιπόν αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να χρηματοδοτηθούν καλύτερα ε, την επόμενη επταετία και έτσι να στηριχθούν περισσότερο. Και ο Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος ε, και να έχουμε σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο καλύτερη συνεργασία όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Το σλόγγαν της χρονιάς πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν «Το παρελθόν συναντάει το μέλλον». Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συνεχής ροή, ότι η κληρονομιά δεν είναι κάτι άψυχο, ότι δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, ε, η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά στρέφεται και στο μέλλον. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια σημαντική δημιουργική βιομηχανία που χρησιμοποιεί τις ζωογόνους δυνάμεις της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και υπάρχουν και κοινότητες ε, για τις οποίες η πολιτιστική κληρονομιά είναι πραγματικά ε, μια δύναμη για να μπορέσουν να επιβιώσουν στους, σε δύσκολους καιρούς, να ανοίξουν τις πόρτες τους σε νέες κοινότητες και να βρουν εταίρος σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Αυτό που προσπάθησα να κάνω πέρσι και που συνεχίζεται και φέτος είναι μια καταγραφή των ευκαιριών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας από κάτω προς τα πάνω. γιατί νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο, αν δηλαδή αποφασίζουμε σε ανώτατο επίπεδο και επιβάλλουμε τις αποφάσεις προς τα κάτω στους πολίτες, νομίζω ότι αυτό το μοντέλο δεν θα είναι βιώσιμο. Αν όμως μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, ξεκινώντας σε τοπικό επίπεδο, όπως ε, και το έρασμος άλλωστε, που βασίζεται στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, στην προσωπική εμπειρία, στην ανάπτυξη δικτύων, επικεντρώνεται στις νέες γενιές. Και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ενισχύεται επίσης και από το ευρωπαϊκό έτος. Και όλα αυτά μετά αντανακλώνται στις προσωπικές σχέσεις. Ναι, μα κατά αυτόν τον τρόπο αναβιώνουμε αυτή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ναυρατίτς. Είναι πολύ ευτυχής που μπορώ να σας συναντήσω εδώ. Συγχαρητήρια γιατί ολοκληρώσατε μια πάρα πολύ έντονη περίοδο εργασιών εγώ ήμουν παρούσα στον τομέα αυτό όταν κάνατε τα πρώτα σας βήματα και σας παρακολούθησα στην προσωπική σας σταδιοδρομία στον τομέα του πολιτισμού και της ε, παιδείας. Έχω δύο ερωτήσεις που έχουν άμεση σχέση με τη θητεία σας. Τον 2018 τον Ιανουάριο οι Υπουργοί Πολιτισμού υιοθέτησαν την δήλωση που έκανε μια έκκληση για τη στήριξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας από τους εταίρους αυτής της διαδικασίας. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει άμεση σχέση με τις ε, δύσκολες ε, συνθήκες που ξεκινήσατε τις εργασίες σας. Θυμάστε το 2015 την χρηματοδότηση, την πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές δομές. Και φτάσαμε σε κάποιους συμβιβασμούς και καταφέραμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία, στους κανόνες, στους κανονισμούς όσον αφορά την στήριξη των υποδομών του πολιτισμού. Τα πράγματα δεν είναι βεβαίως σήμερα ρόδινα όσον αφορά τη χρηματοδότηση του πολιτισμού. Εσείς τι αφήνετε πίσω σας, αφήσατε νομίζετε περισσότερα αποτελέσματα, περισσότερες μελέτες που δείχνουν ότι οι επενδύσεις στην υποδομή του πολιτισμού συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, ότι υπάρχει δηλαδή θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την ανάπτυξη όταν επενδύουμε στις υποδομές του πολιτισμού. Ευχαριστώ και εγώ σας συγχαίρω για την επανεκλογή σας. Να ξεκινήσαμε μαζί. Ήσασταν τότε στο Υπουργείο όταν ξεκίνησα εγώ σαν Επίτροπος και θυμάμαι πολύ καλά την πρωτοβουλία της Λετωνίας για την εβδομάδα του δημιουργικού τομέα και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Τώρα για το μέλλον τι θα αφήσω στον ε, επίτροπο που θα με διαδεχθεί καινοτομία και πραγματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το υποβάλει αυτό σαν πρόταση όπως και πολλά άλλα χρήσιμα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διακήρυξη του Νταβός είναι κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, από θεωρητικής απόψεως, η διακήρυξη του Νταβό συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερες χώρες από αυτές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεπερνάει δηλαδή τα δικά μας σύνορα, αλλά φυσικά και στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Στηρίζουμε τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο συμμετέχει σε αυτήν την πρωτοβουλία. Η υπογράμμιση της σημασίας του πολιτισμού σε τέτοιο υψηλό επίπεδο λήψης αποφάσεων είναι κάτι το εξαιρετικά θετικό. Πολύ καλή ιδέα. Και εννοείται ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε στο μέλλον. Όσον αφορά τα ανώτατα όρια για τις επενδύσεις στον τομέα του πολιτισμού, εγώ τότε είχα προσπαθήσει να πείσω την συνάδελφο Κορίνα Κρέτσου, την επίτροπο Κορίνα Κρέτσου, για να αυξηθούν οι επενδύσεις και μάλιστα σας είχα ζητήσει τότε να στείλετε επιστολές, δημιουργήσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο λόμπι για να πιέσουμε την κυρία Κρέτσου και κάτι πετύχαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε και όταν προετοιμάζαμε τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου του επόμενου, είδαμε περισσότερες συγκλήσεις και θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να χειριστούμε όλες αυτές τις δυνατότητες χρηματοδότησης είτε από ευρωπαϊκά είτε από περιφερειακά κονδύλια. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων, την διακυβέρνηση της χρηματοδότησης και ότι τέτοιου είδους δυσκολίες και προβλήματα θα εξαλειφθούν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσον έχει το λόγο, συντονίστρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την παρουσίαση. Είχαμε σίγουρα πολύ καλή συνεργασία μαζί σας. Αυτό φαίνεται, αν και είμαι νέο μέλος, το διαπιστώνω. Το θέμα της ψηφιοποίησης της κοινωνίας, η οποία διαρκώς αυξάνεται αύριο το πρωί, θα συζητήσουμε πάλι το θέμα αυτό. Το ίδιο α, συζητήσαμε και σήμερα, η ενίσχυση αυτής της α, ψηφιοποίησης το θέμα της αύξησης της χρήσης των ε, κοινωνικών μέσων, τα πλήγματα στην ε, πνευματική και ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων, πώς θα στρέψουμε τους νέους μας και τα παιδιά προς περισσότερη άσκηση, περισσότερο αθλητισμό. Και την ίδια ώρα τα μαζικά φαινόμενα των ε, εικονικών αθλημάτων, e-sports, ηλεκτρονικά σπορ, αυτό είναι κάτι που βεβαίως κατευθύνεται από τον τομέα αυτό των ε, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και είναι κάτι που δια, διαρκώς ε, αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Πίσω από όλο αυτό το τομέα βεβαίως βρίσκεται το κέρδος. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτά τα αρνητικά φαινόμενα, τα οποία είναι αλληλένδετα με την ψηφιοποίηση, πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά μας, έτσι ώστε να συνεχίσουν να βλέπουν τον όμορφο κόσμο μας και να μην είναι μονίμως μπροστά από μια οθόνη. Πώς μπορούμε να δώσουμε λοιπόν κίνητρα και να κινητοποιήσουμε μια στροφή των νέων προς άλλες κατευθύνσεις. I would go Θα ήθελα να πω μικρότερα το εξή. Εμένα δεν με ενθουσιάζουν αυτά τα e-sports. Ακόμη και το όνομα ε, μπορεί να μας οδηγεί σε λανθασμένες ε, αντιλήψεις. Δεν υπάρχει σπορ, αθλητισμός, μόνο το e υπάρχει. Πρόκειται για μία πολύπλοκη δράση. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί επίτροποι εργάζονται ο καθένας στην, στον τομέα του για να μπορέσουμε όλοι να καταλήξουμε σε, μια, σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν μιλάμε μόνο για καλή διατροφή, για καλή άθληση, για ευημερία, αλλά όλα αυτά μαζί. Συν εκπαίδευση και συνδυασμό όλων. Νομίζω ότι οι προκλήσεις στο μέλλον θα είναι ακόμη πιο πολύπλοκος. Η παχυσαρκία, πίν στι διάφορες κοινωνίες ή τα εκπαιδευτικά προβλήματα ή η κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλισμός. Είναι προβλήματα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε ώστε να καταλήξουμε σε λύσεις και καλά αποτελέσματα, διότι η κάθε πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να έχει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα. Αν μιλήσουμε μόνο για εκπαίδευση, χωρίς να λάβουμε υπόψη τον αθλητισμό, την άθληση, το πολιτιστικό, ε, αν θέλετε, πρόσημο, δεν κάνουμε μόνη, από τίποτα. Πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα και θα πρέπει όλες αυτές οι πολιτικές να αποτελέσουν ε, έναν ε, διαδραστικό, αν θέλετε, σύνολο με τον οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος, ακόμη και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως Επίτροπος. Είναι δύσκολο να προσελκύσει κανείς ε, τους νέους σε διάφορους το τη ζωή, στην καθημερινότητα. Θα πρέπει από κοινού λοιπόν να αφιερώσουμε προσπάθειες. Ολοκληρώσαμε με τον ε, γύρο των συντονιστών. Μπορούμε τώρα να παίρνουμε τις ερωτήσεις 2-2. Περιοριστείτε παρακαλώ πολύ σε ένα λεπτό. Ο κύριος Έλερ παίρνει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση. Το θέμα της έρευνας. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες εδώ και πολύ συγκεκριμένες ε, συμβάσεις ε, απορρέουν από τον τομέα αυτό. Δεν έχει βεβαίως αποφασιστεί κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον ε, ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας αλλά και εδώ υπάρχουν θέματα διακυβέρνησης. Μιλήσατε πολύ προσεκτικά για το θέμα αυτό, λέγοντας ότι υπάρχει συνεργασία, ότι υπάρχει συντονισμός. Εγώ θα μιλούσα για διακυβέρνηση. Γιατί κάποια από αυτά που προσπαθήσαμε να κάνουμε αποτύχανε. Γιατί. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και με ευχαρίστηση άκουσα ότι εστιάζετε, εστιάζετε την προσοχή σας στους νέους και πόσα πολλά νέα παιδιά εσείς συναντήσατε. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω όταν τον Οκτώβριο θα καλέσω νέα παιδιά, κυρίως παιδιά τα οποία παρακολουθούν μαθήματα επαγγελματική κατάρτισης και μαθητείας, να τα συναντήσετε. Ξέρω ότι θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας και θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για το με ποιο τρόπο μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα νέα παιδιά για το μέλλον. Um, two tough questions. <laughs> Πολύ, πολύ δύσκολες ερωτήσεις μου κάνατε. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα της, ε, ε, του μοντέλου διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Ε, εξετάζουμε και τα θέματα της νομοθεσίας για το μέλλον και έχουμε έρθει σε επαφή με τα κράτη-μέλη και πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα. Πρώτα απ' όλα το θέμα της αριστείας και δεύτερο το θέμα τη γεωγραφικού ισοσκελισμού. Όταν μιλούμε για διακυβέρνηση λοιπόν στους τομείς αυτούς, αυτοί οι δύο πυλώνε μπορεί να είναι προφανεί για μας, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μιλούμε για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Εγώ δεν θα το έλεγα διακυβέρνηση, αλλά θα έλεγα πώς θα βρούμε ένα σύστημα να επηρεάσουμε τα πράγματα, ώστε να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, διότι τα κονδύλια είναι σημαντικά και έχουμε περισσότερα κονδύλια για το Εράσμους σήμερα. Αν μπορούν να διπλασιαστούν ή να τριπλασιαστούν, αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερα κονδύλια για τα πανεπιστήμια. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Τα πανεπιστήμια έχουν την εντύπωση, αισθάνονται ότι υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο ανταγωνισμό. Έχουμε πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Δυστυχώς, εάν δούμε την, ε, την ταξινόμηση αριστείας, θα δούμε ότι τα, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία είναι τα πρώτα, είναι τα αγγλικά, βεβαίως το πολυτεχνείο το γερμανικό και τα πολυτεχνία της Ελβετίας είναι στις καλύτερες, θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρουμε ότι έχουν μεγάλες επιτυχίες στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Έχουμε 17 συμπράξεις, συμμαχίες αν θέλετε. έχουμε στο τέλος του έτους θα δημοσιεύσουμε κάποια σχετικά γραφά και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αν υπάρχουν προβλήματα θα θέλουμε να τα διορθώσουμε για την επόμενη χρονιά. Απ' την άλλη, δεν μπορεί κανείς να επηρεάσει τα πανεπιστήμια. Βεβαίως, σεβόμεθα απολύτω την αρχή της ανεξαρτησία τους, αλλά μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ επικοδομητική εταίρη. Και στον τομέα της έρευνας θα είχαμε και μία πάρα πολύ καλή λύση και δεδομένου ότι στα πανεπιστήμια πάντα ε, τονίζεται η σημασία των ερευνητικών κέντρων και της έρευνας. Ίσως λοιπόν Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και η εκπαίδευση θα ήταν σίγουρα ο πιο επιτυχής τομέας συνεργασίας. Τι ενθαρρυντικό μήνυμα θα μπορούσα να δώσω στους νέους. Κατά την άποψή μου είναι πολύ θαραλέα άτομα οι νέοι. Διότι κάνουν ό,τι θέλουν αλλά πολλές φορές δεν απολαμβάνουν αυτά το οποία ήθελα να Έχουμε πρόβλημα γύρανσης στην Ευρώπη. Έχουμε γυράσκουσες ε, ε, χώρες. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι καλό. Θα μπορούσε να είναι η λύση για το μέλλον. Τα τελευταία πέντε χρόνια Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι βρίσκεται και συλλογικά και ατομικά στην εκπαίδευση. Όσο περισσότερο εκπαιδευμένη μια κοινωνία, τόσο περισσότερο έχει δυνατότητες ανάπτυξης στο μέλλον. Ελπίζω λοιπόν ότι η εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει σε πιο συνεκτικές κοινωνίες. Άρα θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά εκπαιδευτικά συστήματα για τους νέους και για πολύ άλλο κόσμο που θέλει περαιτέρω στην κοινωνία να προοδεύσει. Ευχαριστώ. Οι δύο επόμενες ερωτήσεις. Thank you for, for the floor, Madam Chair. And I will switch to Hungarian, <laughs> to our common uh, language. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω στα Ουγγαρικά. Köszönni ezt a közösen eltöltött évet, nekem is, mint Nagyon jó volt. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ καλά αυτά τα πέντε χρόνια συνεργασίες και είναι εξαιρετικό το ότι είχαμε έναν Ούγγρο ε, επίτροπο που ασχολήθηκε με αυτά τα πολιτιστικά θέματα. Ήταν λοιπόν πέντε χρόνια πολύ θετικά, επικοδομητικά. Μπορέσαμε να ενισχύσουμε πάρα πολλά προγράμματα που τέθηκαν σε κίνηση το παρελθόν και τώρα βλέπουμε ότι προχωρούν όπως το Erasmus Plus και πάρα πολύ ε, θετικό ήταν το ότι παρακολουθήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία και τις εξελίξεις και δημιουργήσαμε για θέματα πολιτιστικά ένα τόσο ε, θετικό κλίμα. Χαίρομαι που μπορέσατε κι εσείς να ασχοληθείτε με θέματα τόσο λεπτά και ευαίσθητα, όπως αυτό των ακαδημαϊκών τίτλων. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις ε, κοινωνίες μας. Τα θέματα τα πολυπολιτισμικά, της πολυγλωσσίας της διάφορες κοινωνίες μας σήμερα που είναι διαφορετικές από το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Επίσης ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλά υπέρ της κουλτούρας της Ουγγαρίας και της γλώσσας μας. Διότι ξέρουμε ότι η κατάσταση πολιτική είναι πολύπλοκη και ελπίζω ότι ο επόμενος επίτροπος θα σας νοιάζει σε αυτά που κάνει. Θα συνεχίσει την εργασία σας και η συνεργασία μας θα είναι αγαστή. Σας ευχαριστούμε και πάλι και καλή επιτυχία στο μέλλον κύριε Επίτροπε. Ε, ε, Ο κύριος Νίνας, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ σήμερα. Οι άλλοι σας ήξεραν για πέντε χρόνια, σας είχαν γνωρίσει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είμαι λίγο μπερδεμένο, γιατί από τη μια λέτε ότι θέλετε να στηρίξετε τη νεολαία, να τους δώσετε μέσα και από την άλλη λέτε ότι τα ηλεκτρονικά αθλήματα δεν είναι αθλήματα. Εγώ θα πρέπει να τονίσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την, τον πολιτισμό των νέων, την κουλτούρα των νέων, είναι αθλήματα. Ας, ε, για παράδειγμα, η Φόρμουλα 1. Ας δείτε το σκάκι, ένα άλλο παράδειγμα. Πόσοι ασχολούνται με αυτό ηλεκτρονικά. Και θα ήθελα να σας πω, ε, δεν είναι μόνο γιατί θέλω να σας πω κάτι καινούριο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την, τα ευρωπαϊκά αθλήματα και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά γενικότερα και για τον αθλητισμό. Να μπορέσει να αποδεχτεί το γεγονό ότι τα ηλεκτρονικά αθλήματα είναι πλέον μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια τεράστια επιχειρηματικότητα πίσω από αυτά και πίσω από τα βίντεο παιχνίδια. Και θα πρέπει αυτό να το αποδεχτούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολύ σημαντικές επιχειρήσεις στη Γερμανία, την Πολωνία. Υπάρχει το Select Project Red και υπάρχουν και οι προγραμματιστές στον τομέα αυτό. Δημιουργούνται λοιπόν θέσεις εργασίας, είναι σημαντικός ο κλάδος και ήθελα να το τονίσω. Πρέπει να τους ενισχύσουμε. Επίσης, το ηλεκτρονικά αθλήματα είναι ε, ένας δρόμος για να φτάσουν οι νέοι στα πραγματικά φυσικά αθλήματα. Και Βεβαίω ξέρουμε ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή είπε ότι ναι, δεν ε, είναι αθλήματα, δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά δεν είναι αλήθεια. Τα ηλεκτρολικά αθλήματα ε, ενισχύονται όλο και περισσότερο και είναι σήμερα πολύ πιο σημαντικά από ότι είναι η Ολυμπιακή αγώνες. Μαζί λοιπόν με τον κλασικό αθλητισμό θα πρέπει να αναπτύξουμε και τον ηλεκτρονικό αθλητισμό. Σας παρακαλώ λοιπόν τις υπόλοιπες εβδομάδες που θα είστε ακόμα επίτροπος να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας για να μπορέσετε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Βλέπω τα πρόσωπά σας, ξέρω ότι δεν συμφωνείτε όλοι. Ε, δεν μπορούμε όλα βεβαίως να τα προβλέψουμε αλλά για τους νέους ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ακούμε τις διαφορετικές απόψεις. Μιλήσαμε όμως για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών που περνάνε τις μέρες τους, ολόκληρες μέρες μπροστά από το διαδίκτυο, μπροστά από μια ε, οθόνη και δεν κάνουν κανένα ε, σωματικό, καμία σωματική άσκηση. Για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε. Άλλο είναι αν θέλετε το να κοιτάει κανείς και να παίζει ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό που αφορά τη Φόρμουλα 1 και άλλο να μπει μέσα στο όχημα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα, αν συγκρίνετε, αν θέλετε, το θέμα της συγκέντρωσης, η συγκέντρωση όταν κάποιος παίζει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι τεράστια. Άλλο λέω εγώ, λέει η πρόεδρος, δεν μίλησα για συγκέντρωση, μίλησα για σωματική άσκηση. Δεν συγκρίνεται ένας που οδηγεί μια Φόρμουλα 1 και ένας που παίζει το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αυτό είπα. Ε, Ουσιαστικά συμφωνούμε. Συμφωνώ και εγώ, αλλά από την άλλη είμαι υπεύθυνο για τον αθλητισμό και όχι για την ε, επιχειρηματικότητα. Όταν λοιπόν μιλάω για αθλητισμό, αναφέρομαι σε κάποιες αρχές. Πρώτα-πρώτα, την ε, σωματική δραστηριότητα. Μετά, τον, την, μια συμπεριληπτική κοινωνία και δραστηριότητες για τους πολίτες. Τα ηλεκτρονικά αθλήματα δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Μπορεί να υπάρχει μια άνθηση του κλάδου, μπορεί να είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός τομέας, ε, δεν αντιλέγω, αλλά Νομίζω ότι ε, κάθε δραστηριότητα των πολιτών και κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με την ε, φυσική δραστηριότητα δεν πρέπει να συγχέεται με τα ηλεκτρονικά χρήματα για τα οποία δεν θα ήθελα να δοθεί χρηματοδότηση. Εγώ συγκεντρώνομαι σε αυτά που είναι τα παραδοσιακά αθλήματα, με την φυσική άσκηση, με τη φυσική δραστηριότητα. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανείς καθισμένο στην καρέκλα του, θα έλεγα. Το σκάκι που είπατε, εγώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε από ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που μπορούμε όμως είναι να ενισχύσουμε δραστηριότητες πολιτών που χρειάζονται χρηματοδότηση και που δίνουν στους πολίτες την χαρά, την εμπειρία της πραγματικής κίνησης, του να κινούνται με το σώμα τους. Ο κύριος Φραγκόφσκι και η Τζούλι Βόρντ έχουν το λόγο. Jak jesteśmy już przy sporcie, to i może chwilę pozostańmy μιλάμε για αθλητισμό. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Ήταν μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής, ήταν μια πρωτοβουλία η εβδομάδα του αθλητισμού. Ποιες όμως είναι οι δυνατότητες επικύρωσης της συμφωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά τον αθλητισμό εκ μέρους των κρατών μελών. Επίσης, το θέμα της επικύρωσης εκ μέρους τρίτων χωρών. Διότι υπάρχουν τρίτες χώρες που δεν έχουν επικυρώσει συμφωνίες. Και εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Με συγχωρείτε. Για τους συναδέλφους που φεύγουν. Έχω να πω κάτι για τον αθλητισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί όσον αφορά τον ορισμό του πολιτισμού. Αυτή θα πρέπει να είναι η θέση μας. Εμείς διαμορφώνουμε πολιτική που έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Για μένα η τέχνη του δρόμου, η street art, είναι μια πάρα πολύ σημαντική μορφή τέχνης. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ, να οργανώσουμε ε, μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την ε, τέχνη του δρόμου. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, γιατί οι νέοι είναι που φτιάχνουν τον πολιτισμό, που δημιουργούν τις νέες μορφές πολιτισμού. Δεν είναι εγκλωβισμένοι από τον δικό μας ορισμό του πολιτισμού. Και νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να διαβρύνουμε την προοπτική μας υπάρχουν μερικοί που θεωρούν ότι τα γραφίτι δεν είναι μορφή τέχνης. Αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτούς τους νέους ορισμούς, τις νέες μορφές τέχνης. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές τέχνης, οι οποίες μάλιστα ε, συνδυάζονται μεταξύ τους, μπερδεύονται. Είναι, παίρνουν κάτι από εδώ, παίρνουν κάτι από εκεί, κάτι από την κληρονομιά και το ανακυκλώνουν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτές τις νέες μορφές τέχνης. Αυτά. Συμμετείχα λοιπόν στους ειδικού Ολυμπιακούς στο Λονδίνο, τους παραολυμπιακούς, συγγνώμη, στο Λονδίνο και ήταν ε, μια πραγματική εμπειρία για μένα, γιατί δεν ήταν ανάγκη να τρέξεις, μπορούσες και να περπατήσεις και να χορέψεις και να πηδήξεις και να πας αναπηρικό καροτσάκι και ήταν πολύ σημαντικό να συμμετείχω μαζί με τους άλλους. Το σημαντικό δεν ήταν να κερδίσει κανείς, αλλά να έχει αυτή την αίσθηση ότι κάτι πέτυχε. Αυτό. Και έχω να πω και κάτι άλλο. Εσείς θα φύγετε κύριε Επίτροπε, αλλά στο επιτελείο σας, ε, στην Επιτροπή υπάρχουν ε, πολλά αξιόλογα άτομα. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για μας ε, η συζήτηση μαζί τους και ε, ε, βεβαίως και η κριτική που ασκήσαμε, αυτός είναι ο ρόλος μας. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρετε στο επιτελείο σας την εκτίμησή μου και ε, πόσο εκτιμούμε τη συνεργασία τους μαζί μας. Νομίζω ότι κάποιοι λοιπόν θα ασχοληθούν με το νέο θεματολόγιο για την εκπαίδευση. Ε, δεν ακούσαμε όμως κάτι για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του τύπου. Ίσως πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο στο θεματολόγιο. Μπορείτε να το μεταφέρετε αυτό στο επιτελείο σας. Μπορούμε να συνεργαστούμε γι' αυτό. Και θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την στήριξή σας για την ε, έκθεση που είχα κάνει όσον αφορά τον ε, ε, διάλογο, τον διαπολιτιστικό διάλογο και το πώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να διδαχτεί και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να, ε, μπορούμε να τον διευκολύνουμε ε, μέσα στις ε, σημερινές κοινωνίες. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να συνεχιστεί, για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι και εδώ μιλάω για την για την ε, πολιτιστική διπλωμασία, διπλωματία, διότι σκοπός της είναι να ε, προλάβει τις ε, συγκρούσεις, να προωθήσει την ειρήνη και εδώ βέβαια σκέφτομαι το πρόβλημα των, το προσφυγικό και επίσης εσείς διαθέσατε την ανάλογη χρηματοδότηση, ήταν πολύ σημαντικό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Κοιτάξτε, θέλω να δώσω λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει. Μην μιλάτε κάθε φορά δύο λεπτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ο κύριος Γεωργούλης έχει το λόγο. Τώρα δουλεύει προφανώς, ε. Κύριε Επίτροπε, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα ε, ομιλία σας ε, σήμερα και θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτού του είδους ο διάλογος και κυρίως όταν φτάνουμε σε πρακτικές όπου είναι φυσικά ε, δυνατόν. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με ε, το 25ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνού Συμβουλίου ε, Μουσείων που γίνεται αυτές τις μέρες στο Κιώτο της Ιαπωνίας. Το βασικό αντικείμενο της ε, συζήτησης στο συνέδριο αυτό είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας και της ταυτότητας των σύγχρονων μουσείων. Ε, πέρα από λαμπρές ε, εξαιρεσει. τα μουσεία έχουν ουσιαστικά εγκλωβιστεί στο παρελθόν τους και μας, ε, τους έχουν πιάσει μια ισοστρέφεια. Ε, αντί να είναι φορείς ε, ε, πληροφοριών και να συμβάλλουν στα βασικά θέματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο, όπως είναι η κλιματική κρίση, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στην παιδεία, πολύ πιο στεναρά. Ε, αντί για να ασχολούνται με αυτά, εγκλωβίζονται στο παρελθόν τους. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν προφανώς ξέρετε την, το συνέδριο αυτό, Εάν η Κομισιόν ε, παίρνει θέση απέναντι στους καινούργιους όρους, αν έχει ε, σκοπό να συμβάλλει σε κάποια αλλαγή και κάποια βελτίωση αυτού του όρου και τι ενέργειες θα, ήθελε, θα έχει στην ατζέντα της για το μέλλον πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πληροφορίες για τη διάσκεψη την οποία αναφέρατε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι η παράνομη διακίνηση έργων τέχνης είναι κάτι το οποίο μας στερεί εμάς από αυτά τα έργα, τα αριστουργήματα και είναι κάτι το οποίο το συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρχει μια σχετική νομοθεσία. Αυτό αφορά το παρόν. Τώρα, το τι έγινε στο παρελθόν είναι θέμα διμερών ρυθμίσεων και διαπραγματεύσεων. Στη Γερμανία, Φερρυπίν, όπως και στη Γαλλία, γίνεται συζήτηση για το πώς θα επανέλθουν κάποια έργα τέχνης που βρίσκονται στα μουσεία στις χώρες που ανήκουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα δεν έχει λάβει θέση για τέτοιου θέματα διότι δεν υπάρχει και η νομική βάση για κάτι τέτοιο. As for the, uh, for the arts and refugees... Τώρα, για την uh, θέμα των προσφύγων, της δημιουργικότητά τους στα και για τα πολιτιστικά θέματα και η κουλτούρα δεν είναι για μένα μόνο κάτι το οποίο κάνει κανείς για να ψυχαγωγηθεί. είναι μέρος της κουλτούρας μας και το Creative Europe νομίζω ότι μπορεί να παίξει όπως και το Εράσμου ρόλο στον κοινωνικό, στην κοινωνική συμπερίληψη κάποιων ατόμων στις κοινωνίες μας. Πρόκειται για κάτι το οποίο γίνεται τώρα και θα αποφέρει καρπούς στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική συμπερίληψη κάποιων ατόμων. Ευχαριστώ. Υπάρχει και άλλη ερώτηση από τον κύριο Γεωργούλη, συμπληρωματική. I think that we got, uh, we got lost in translation. Uh, didn't mean what's going on with uh, museums right now. I mean that... Um, Νομίζω ότι χαθήκαμε στη μετάφραση. Δεν εννοούσα κάτι που συμβαίνει στη μετάφραση τώρα. Να συνεχίσω στα ελληνικά. Ε, ο ορισμός πρόκειται να επαναπροσδιοριστεί. Όχι το μουσείο σαν ε, μουσείο. Αυτό εννοούσα στο, στον προηγούμενο λόγο που έκανα. Ε, στο 25ο Παγκόσμιο Συνέδριο ο, θα πρόκειται να συζητήσουν για τον επαναπροσδιορισμό του ορισμού της έννοιας μουσείου και της ταυτότητάς του. Τι ακριβώς είναι το μουσείο και τι ακριβώς προσφέρει στον κόσμο. Και αν η Κομισιόν πάνω στο θέμα αυτό έχει ε, άποψη, φαντάζομαι θα έχει μία άποψη, και εάν πρόκειται να συμβάλλει σε αυτή την, ε, την αλλαγή για παράδειγμα υπάρχουν μουσεία τα οποία ε, ας, τα πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση νεκρά μουσεία δηλαδή υπάρχουν τα εκθέματα από το παρελθόν και είναι μόνο αυτό έρχεται ο επισκέπτης, βλέπει το μουσείο, καταλαβαίνει τι είναι το έκθεμα, καταλαβαίνει τι γίνεται από την ιστορία, τον καλλιτέχνη και όλα αυτά και το παίρνει στο μυαλό του όλο αυτό και υπάρχουν τα open museums αυτή τη στιγμή που μπορεί ο επισκέπτης να επισκεφθεί και να ζήσει την εποχή, όχι απλώς να τη δει από απόσταση, να γίνει μέρος αυτής της, ε, της ε, ε, αυτού του εκθέματος. Ε, κάπως έτσι πιστεύω ότι πρόκειται να αλλάξει και ο ορισμός και αν η Κομισιόν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την αλλαγή και να δημιουργήσει και νέες γραμμές ίσως, ώστε οι άνθρωποι που θα πηγαίνουν στο μουσείο να μην είναι απλώς επισκέπτες, αλλά να γίνονται μέρη του εκθέματος και ίσως αυτό εκπαιδευτικά να έχει ακόμα και πιο βαθύ ε, αντίκτυπο στον κόσμο. Well, frankly, I'm not sure if the... Δεν ξέρω αν η κοινότητα των επαγγελματιών θα δει με θετικό μάτι την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επατροπής. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ κακή εμπειρία όσον αφορά τέτοιου είδους ε, προτάσεις. Ας αφήσουμε τα μουσεία, ας αφήσουμε την διατύπωση του μέλλοντος των μουσείων στα χέρια των επαγγελματιών, γιατί δεν είμαι, αν θέλετε, ειδικό, καθόλου ειδικό στα θέματα αυτά. Είμαι αρμόδιος για πολιτιστικά θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ειδικό θέμα και ας αφήσουμε τους επαγγελματίες να το χειριστούν. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επίτροπο για την πενταετία που συνεργαστήκαμε, για τη στήριξη που παρήχε στις δικές μας ιδέες και τις πρωτοβουλίες μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα εσείς μας προτείνατε. Πολλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα πρέπει να συνεχιστούν, να εξελιχθούν και πιστεύω ότι μιλάω εδώ εκ μέρους όλες της Επιτροπής και για την εκπαίδευση και για τον πολιτισμό και για τον αθλητισμό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και για εξυγχρονισμό αλλά και για καλύτερη χρηματοδότηση. Πραγματικά νομίζω ότι η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των ευρωπαϊκών λαών δεν μπορεί παρά να περάσει από κάτι τέτοιο και φυσικά ο αθλητισμός εδώ πρέπει και μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο και όταν λέω αθλητισμό εννοώ σωματική άσκηση. Στο παρελθόν λοιπόν η συνεργασία μεταξύ ημών ήταν εξαιρετική, ελπίζω να ανανεωθεί. Αν δεν σας ξαναδώ, σας εύχομαι κάθε καλό και σας ευχαριστώ πραγματικά για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αύριο το πρωί παρακαλώ να είστε στην ώρα σας, ακριβώς 9, για να συνεχίσουμε. Αύριο το πρωί επίσης θα έχουμε συνάντηση των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.